Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Να σας ε, ενημερώσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ακούγομαι. Ωραία. Πρέπει να μιλάω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τη... Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σας έχει διανομηθεί στις 11 Απριλίου του 2011 και σας προτείνω να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη δύο νέα σημεία. Καταρχάς, είχα ένα αίτημα του Υπουργού Οικονομίας ε, Τζούλιο Τρεμόντι της Ιταλίας να έρθει εδώ στην Επιτροπή να μιλήσει για θέματα τα οποία αφορούν την οικονομική κρίση, αλλά πιο συγκεκριμένα τη χρηματοοικονομική κρίση και το θέμα τα μετανάστευση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και τα θέματα ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαένων πρόσωπο και ζήτησα από τους αδέλφους ε, του ΕΛΚΑ, ε, από τους φιλελευθέρους και τους σοσιαλιστές. Δεν μου είπε κάποιος ότι έχει αντίρρηση, επομένως θα ήθελα να προσθέσουμε το σημείο αυτό ε, στις 11.30 αύριο το πρωί. Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσουμε και την έκθεση ε, συγγνώμη, τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, με συντάκτη τον κύριο Μέσερ Σμιτ και θα το συζητήσουμε σήμερα στις 18 Απριλίου για την καλύτερη νομοθεσία είναι η γνωμοδότηση και θα πρέπει να γίνει πριν από τις συνεδρίες των συντονιστών. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας εγκαίρως στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω δύο νέα μέλη, αναπληρωτές, η κυρία Σουζάνα Μπροτσποχάτα, ελπίζω να πρόφερα καλά το όνομά σας, δεν είναι εδώ, ε. Και τον κύριο Τζον Στρουετ Αγνιού, ο οποίος επίσης δεν είναι καλά. Ελπίζω να το πρόφερα και αυτό σωστά. Σα έδωσα λοιπόν όλε τι πληροφορίε. Θεωρώ εγκριθήσα την ημερήσια διάταξη με τι τροποποίησεις που σα ανέφερα. Πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά από τι προηγούμενε συνεδριάσει τη 7 η Μαρτίου και τη συνεδρίαση τη 14 και 15 Μαρτίου. Έχετε τα πρακτικά στη διάθεσή σα και εάν δεν υπάρξουν ενστάσει και παρατηρήσει, ε, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Δεν βλέπω κάποιον να έχει ενστάσει. Ωραία, να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη εξελίξεις στην Κοζάκ. Είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος Μικέλ Άγχελ Μαρτίνες Μαρτίνες. Τον καλωσορίζουμε. Έχει άλλωστε έρθει επανειλημμένο στην Επιτροπή μας. Θα μπορούσαμε να το θεωρούμε και επίτιμο μέλος της Επιτροπής μας. Και μάλιστα είχε ξαναέρθει και στις 31 Ιανουαρίου και είναι εδώ για μια περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ η οποία θα γίνει ε, στη Βουδαπέστη 29 με 31 Μαΐου. Στόχος τη συνάντηση αυτή είναι να προετοιμαστούμε καταλήλω και να κάνουμε τι κατάλληλε προτάσει ώστε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μεταβεί στη Βουδαπέστη στι 29 ε, Μαΐου να μπορεί να διεξάγει τα καθήκοντά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι αρκετά. Υπάρχει η αξιολόγηση της ε, Ουγγρικής Προεδρίας, το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης, η Ευρώπη 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες τεχνικές τροποποίησεις στον κανονισμό της ΚΟΖΑΚ και επίσης πρέπει και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να μας πει πρωτίστως ο πρόεδρος ε, Μαρτίνεθ μεταξύ άλλων πέρα από κάποιες ε, κατευθυντήρες γραμμές για την επόμενη συνεδρία της ΚΟΖΑΚ να μας πει και τι θα γίνει στην επόμενη διάσκεψη των προέδρων των ε, κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συμμετείχε με τον πρόεδρο Μπούζεκ στις 4 και 5 Απριλίου Συζητήθηκε πολύ και το θέμα της ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ε, εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμενης και για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι, συγγνώμη, νομίζω ότι σας έχουν διανεμηθεί αντίγραφα με τα συμπεράσματα της Προεδρίας και να δώσω απευθεία το λόγο στον πρόεδρο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, τον οποίο ευχαριστώ εκ νέου για την ε, παρουσία του εδώ. Εγώ, Κάρλο, πρέπει να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχω να απευθυνθώ στους συναδέλφους μιας επιτροπής τόσο εξέχουσας όσο ε, παρούσα. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε στη διάσκεψη της ΚΟΣΑΚ στη Βουδαπέστη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καθοριστικό αυτό να συντονιστούμε κάπως λίγο. Να σταθούμε λίγο στις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ιδιαίτερα μετά τη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που έλαβε χώρα εδώ στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες. Θα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους εδώ παρόντες ότι για να συζητήσουμε αυτό το θέμα πήγα στη διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων, πήγα στο διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και είχαμε και τρεις συνεδριάσεις με τον Πρόεδρο Μπούζεκ και με κάποιους εισηγητές. Διότι πραγματικά η κατάσταση χρειάζεται προβληματισμό πέρι συλλογή και απόφαση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξή. Η διάσκεψη των Προέδρων διοργανώθηκε με τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό από τους Βέλγους, μέλη της Γερουσίας και της Βουλής του Βελγίου πολλά ενδιαφέροντα θέματα μας απασχόλησαν, αλλά κυριάρχησε ένα θέμα. Γιατί μπορεί σε κάποια ζητήματα να γίνανε συζητήσεις έτσι με τη συνήθη σύνηση και φρόνηση όσοι ήθιστε μας απορρόφησε στα τρία τέταρτα ένα και μόνο θέμα ε, αφιερώσαμε πολύ περισσότερο χρόνο από εκείνο που είχαμε προβλέψει. Και αυτό είναι αυτό που ανέφερε και εσύ. Η ε, θέση σε ισχύ συνθήκη της Λισαβόνας υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζεται με τα εθνικά για θέματα ε, ασφάλειας, άμυνας και κοινή εξωτερικής πολιτικής. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της Europol και Eurojust, ε, ασφάλεια, ε, δικαιοσύνη, συνεργασία σε αυτά τα θέματα, αλλά ήταν λιγότερο έντονη η συζήτηση. Εγώ φροντίζω πάντα να μιλάω με μετριοπάθεια, αλλά πρέπει να σας πω ότι επικράτησε μεγάλη ένταση και ε, ήταν δυσάρεστη τελικά η κατάσταση διότι πραγματικά με πάρα πολύ οξύ τρόπο είδαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Βελγικού Κοινοβουλίου με κάποια υποστήριξη των Ιταλών και των Γερμανών σε κάποια στιγμή από τη μια και από την άλλη ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Και ορισμένοι μιλούσαν και οι άλλοι που σιωπούσαν ε, συνενούσαν. Γιατί αυτή η ένταση διότι αυτό αποκλειστικά αφορούσε τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, πώς να το πω, οι επιθέσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να τις χαρακτηρίσω έτσι, οι επικρίσεις προς το Βελγικό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ήταν κριτικές για θέσεις που είχε πάρει το Βελγικό Κοινοβούλιο ε, και επεφύλασε κάποια αξιοπρεπή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες, σε αυτή τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να υπάρχει και μια παρακολούθηση από πλευρά κοινοβουλευτική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Είναι γνωστά τα προηγούμενα στους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής. Η Βελγική Βουλή είχε κάνει μια πρόταση, ένα κείμενο εν πάση περιπτώσει, για το πώς θα μπορούσε να διαρθρωθεί αυτή η συνεργασία και επαναλαμβάνω η συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει ή ε, μας να συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό το έγγραφο του Βελγικού Κοινοβουλίου είχε διαβιβαστεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια ομάδα εργασίας που παρακολουθεί τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και κατέληξε ε, εκεί ότι ήταν ικανοποιητικό αυτό που πρότεινε το Βελγικό Κοινοβούλιο. Είχε μια αρχιτεκτονική διάσκεψη σε αυτό ε, διάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ας πούμε, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, με όρους ενός τρίτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο τρίτα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάθε έξι μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αναλάμβαινε και τη γραμματεία κτλ. Η δική μας ομάδα εργασίας ζήτησε να ανέβουμε από το 33% στο 40%. Η διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων θεώρησε ότι δεν ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Απλώς να στείλουμε μια επιστολή, έλεγε, στο Βελγικό Κοινοβούλιο και να πούμε ότι συμφωνούμε απολύτως με το Βελγικό έγγραφο. Αυτή ήταν η φρόνιμη γραμμή, ας πούμε, η συνετή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια, χωρίς καμία εξαίρεση σχεδόν, είχαμε ιδιαίτερα επικριτικές αντιδράσεις μετά απέναντι στο Βελγικό Κοινοβούλιο ως προς τον τόπο της συνεδρίασης, ως προς τη γραμματεία και κυρίως ως προς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το οικοδόμημα, ας πούμε, σε αυτή την αρχιτεκτονική. Ακολούθησε δεύτερο έγγραφο του Βελγικού Κοινοβουλίου, όπου λέει ότι ε, συντόνισε και συγκέρασε τις διάφορες απόψεις που συνέλεξε. Βασικά τι έκανε, υποβάθμιζε λίγο, αλλά διατηρούσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διατηρούσε ένα 20%. Γιατί είπε ότι, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι φτάνει στο 1 τέταρτο της συμμετοχής, ε, έχοντας το 20% του συνόλου της διάσκεψης, στο 1 τέταρτο των όσων έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ακολούθησε η συνεδρίαση εδώ στις Βρυξέλλες και η κατάσταση πρέπει να σας πω ήταν πάρα πολύ ε, τεταμένη διότι έγινε μια περίεργη συμμαχία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ορισμένα κοινοβούλια που είναι ρητά και κατηγορηματικά αντίθετα ε, με το οτιδήποτε αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε έτσι, υπηρετική αντίληψη για τα πράγματα στην Ευρώπη και αντιδρούσαν σε όλα. Και στην εξωτερική πολιτική και στην κοινή εξωτερική ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας και όλα αυτά, όχι σε όλα. Μαζί με αυτούς όμως εμφανίστηκαν και άλλα κοινοβούλια και ήταν πολύ περισσότεροι εκπρόσωποι που θεωρούσαν ότι αυτό που θα πρέπει να φτιάξουμε δεν είναι ένα δίκυκλο, αλλά ένα 28 κύκλο και ένας τροχός να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 27 τροχή των κρατών μελών. Κάθε κοινοβούλιο να στέλνει μία ρόδα. Γιατί το λέω έτσι. Γιατί αν ενώσουμε ε, ε, όλα τα σώματα όλες τις βουλές φτάνουμε στα 39-40 αλλά εντάξει ε, σε χώρες όπου έχουν κοινοβούλιο με δύο σώματα θα ήταν μία εκπροσώπηση εξού λοιπόν και η ένταση και η οξύτητα που επικράτησε γιατί διαφορούσαμε και διαφέραμε και στην αντίληψη την ίδια μα δεν είναι ορίζει αυτό η συνθήκη της Λισαβόνας και το πρωτόκολλο στα άρθρα 9 και 10, μιλάει πάντα για δύο συνομιλητές. Από τη μια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη τα Εθνικά Κοινοβούλια, όλα μαζί. αλλά ορισμένοι αγνοούν το άρθρο 9 και επικεντρώνονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια στο άρθρο 10, λες και το 9 δεν υπήρχε. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο. Πρώτος πρώτος μίλησε ο πρόεδρος Μπούζεκ και ακριβώς επειδή έχει στο μυαλό του όπως και εμείς αυτό το μέλημα της συνεργασίας και είπε ότι μπορούμε να συμπελάβουμε και μια τελευταία πρόταση του Βελγικού Κοινοβουλίου να έχουμε εμείς λέει 27 εκπροσώπους και τα εθνικά κοινοβούλια 4 έκαστο. Δηλαδή 4 επί 27, 108. Έτσι. 27 εμείς, 108 τα εθνικά κοινοβούλια. Και μετά άρχισε η κολοκυθιά. Όχι 4, λέγανε τα εθνικά κοινοβούλια, έξι να είναι από κάθε κοινοβούλιο. Άρα 27 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 162 από τα εθνικά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πρόθυμος και το είπα να δεχτώ αυτή την ε, πρόταση. Το είχε πει και ο Μπούζεκ ότι το 27 το, συζητάμε, ε, το άλλο που συζητάμε είναι η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και εγώ δεν θα διαφωνούσα δημόσιο με τον πρόεδρό μου. Αλλά μας έκανε έκπληξη το γεγονός ότι μας άρκασαν ως απάντηση. Το μόνο που συζητούσαν που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είμαστε στο 14% πλέον και ούτε αυτό το συζητούσαν. Το μόνο που θέλανε ε, είναι 162 από τα Εθνικά Κοινοβούλια και 6 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας. Οι Βέλγοι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή για να πετύχουν κάτι παραπάνω και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η συνένηση δεν επικράτησε. Και όχι μόνο η συνένεση δεν επικράτησε, αλλά ούτε και για το τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και μπρος. Έγιναν πέντε ή έξι προτάσεις διάφορες και τις απέρριψαν όλες. Η μία πρόταση ήταν η Πολωνική Προεδρία να συγκαλέσει έκτακτη διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων στο δεύτερο εξάμεινο του έτους για να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε. Απερίφθη. Άλλη πρόταση. Δεύτερη, ο πρόεδρος Μπούζεκ και ο πρόεδρος της Πολωνικής Βουλής, που δεν χρειάζεται και διερμηνία, να συνεδριάσουν οι δυο τους για να βρούνε ένα τρόπο να προχωρήσουμε. Απερίφθηκε αυτή η πρόταση. Πρόταση τρίτη. Να συναντηθεί μια τρόικα. Τρεις πρόεδροι των, μεγα... των κοινοβουλίων της Προεδρίας. Η προηγούμενη, η νυν και η επόμενη με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απερίφθη. Και τελευταία πρόταση έσχατη, η Γενική Γραμματή των διαφόρων Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεδριάσουν για να δουν αν μπορούν, ε, εν πάση περιπτώσει, οι υπάλληλοι ε, να ε, λιάνουν το δρόμο που δεν καταφέραμε εμείς οι βουλευτές. Και αυτή απερίφθη. Οπότε μηδέν στο πηλίκο. Καμία απολύτως λύση δεν βρέθηκε για το πώς θα συνεχίσουμε τώρα από εδώ και μπρος. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Οι συζητήσεις που κάναμε με φίλους από την Επιτροπή Εξωτερικών, με τη διάσκεψη των Προέδρων, με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με τον εισηγητή, τον κύριο Ντάφ και τον κύριο Γκουαλτιέρη και τον κύριο Μπρόκ, τους άλλους εισηγητές. Πού καταλήγουμε εμείς, αγαπητοί φίλοι, πρώτον. Αυτό που θα πρέπει να φωτίζει τώρα από εδώ και μπρος τη συμπεριφορά μας είναι η αρετή της υπομονής. Άλλη αρετή που χρειαζόμαστε είναι η καρτερία και η ε, σύνεση. Και δεν χρειάζεται καμία βιασύνη. Εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται καλύτερα και στον τομέα αυτόν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση, ε, ούτε αγωνίες χρειάζονται, ούτε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε ε, φαϊνές ιδέες. Οπότε στα συμπεράσματα που θα έχετε στα χέρια σας, το πραγματικό κείμενο είναι το γαλλικό, που λέει δεν υπήρξε συνένεση για τίποτα. Όχι το αγγλικό κείμενο που λέει ότι δεδομένου, πώς το λέει, ότι δεν συμφωνήσαμε για τίποτα, συμφωνήσαμε, ξέρω εγώ τι διαφοδούμε. Όχι. Είτε εγκρίνονται τα πάντα, είτε δεν εγκρίνεται τίποτα. Έτσι κι αλλιώ πακέτο πάνε αυτά. Πάντω, η σημερινή κατάσταση ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει στα εξή. Πρώτον, να καταλάβουμε ότι χάρη στην εργασία ακριβώς της Επιτροπής σας και άλλων επιτροπών, αυτή τη στιγμή η συνεργασία και η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια λειτουργεί έτσι και αλλιώς, καλώς. Διότι εξορθολογήσαμε μια σειρά πραγμάτων και Έχουμε τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινέ κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Αυτά όλα λειτουργούν θαυμάσια, καλύτερα από το παρελθόν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Εκεί που πάνε στραβά τα πράγματα είναι αυτό που σας είπα και τις προάλλες που είχα μια συζήτηση με τους Πολωνούς συναδέλφους που είχαν έρθει για μια τέτοια μεικτή συνεδρίαση, τους είπα και τους έδωσα δύο εικόνες. Ότι εμείς ας πούμε δύο παρομοιώσεις. Εμείς ε, θέλουμε ένα δίτροχο, αλλά αυτό το δίτροχο δεν θα είναι ένα ποδήλατο του 19ου αιώνα που θυμάστε ότι έχει ένα τεράστιο τροχό 162 εκατοστά διάμετρο και μικρή ροδίτσα να έχει 6 εκατοστά διάμετρο γιατί είναι δύσκολο αυτό το όχημα να προχωρήσει και εξάλλου φάνηκε ε, ότι δεν ήταν χρήσιμο και το στείλαν στα μουσεία της ιστορίας και το αντικατέστησαν από ε, άλλα οχήματα πιο λειτουργικά και πιο χρηστικά. Και η πρόεδρος της Γερουσίας, που είναι πολύ καλή και ευγενική, ε, ε, μας είπε ότι, και της είπα και εγώ, το θέμα είναι και η πρόκληση να μάθουμε να χορεύουμε μαζί. στην αρχή όταν μαθαίνεις να χορεύεις πατάει ο ένας το πόδι του άλλου και τα λοιπά. Μετά όμως μαθαίνεις και ε, χορεύεις σαν ζευγάρι και ακολουθείς και το ρυθμό και τα πάντα. Και αυτή είναι η πρόκληση, να μάθουμε να χορεύουμε. Αλλά ε, χρειάζονται δύο για να θέλουν να μάθουν. Εμείς θέλουμε να χορέψουμε και σφιχτά μάλιστα, αγκαλιασμένοι με τα εθνικά κοινοβούλια. Και είμαστε και υποχρεωμένοι και με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Αυτό όμως θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και εκεί βρισκόμαστε. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε, Κάρλο. Και είναι και ο φίλος μου Μέντες Δεβίγο, ο μάρτυρας. Εγώ διατέλεσα 22 χρόνια εθνικός βουλευτής και 12 είμαι εδώ. Οπότε δεν μπορώ να είμαι ταλιμπάν ούτε ε, για το ένα ούτε για το άλλο κοινοβούλιο. Ούτε ποτέ ήμουν ταλιμπάν, ξέρω εγώ, του σφυριού ή του κατσαβιδιού. Άλλο, άλλη λειτουργία έχει το κατσαβίδι, άλλη λειτουργία έχει το σφυρί. Δεν σημαίνει επειδή είναι εργαλεία ότι πρέπει να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο και τα δύο είναι χρήσιμα και θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ε, με τρόπο αρμονικό και παραπληρωματικό συμπληρωματικό. Λοιπόν, εμείς θα ακολουθήσουμε την πορεία μας, θα δούμε που θα καταλήξουμε, πάντως και τελειώνω με αυτό. Στην Κοσακ, στη Βουδαπέστη, η ημερήσια διάταξη έχει ε, οριστεί όπως ορίζει ο κανονισμός και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τώρα εδώ που φτάσαμε δεν μπορεί να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να ε, εμποδίσει στην αρχή που εγκρίνεται και επίσημα η ημερήσια διάταξη να σηκώθει κάποιο προημερησία διάταξης και να κάνει μια πρόταση η κατάσταση θα είναι περίπλοκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που αυτό που θέλουν είναι η ΚΟΣΑΚ να γίνει μια πλατφόρμα όπου θα συζητείτε και θα παρακολουθείτε η πολιτική ασφαλείας και ε, η ΚΕΠΑ και η ΕΠΑ. Εμάς αυτό δεν μας εξυπηρετεί ούτε το θέλουμε. Το άρθρο 10 λέει, του πρωτοκόλου πάντα, ότι η ΚΟΣΑΚ μπορεί ε, κατά καιρού να συζητάει οποιοδήποτε θέμα θέλει για την εξωτερική πολιτική ή ό,τι άλλο θεωρεί σκόπιμο. Αλλά δεν μπορεί να μετατραπεί ο μηχανισμός εκείνος που με τρόπο συστηματικό και μόνιμο και ε, να είναι το όργανο αναφοράς όπου θα γίνεται ε, αυτό ε, το έργο, αυτή η συνεργασία. Δεν γίνεται αυτό στην ΚΟΣΑΚ. Οπότε στη Βουδαπέστη μπορεί να το βρούμε αυτό μπροστά μα αυτή τη δυσκολία εξού και είναι πολύ σημαντικό, Κάρλο, η αντιπροσωπεία στην ΚΟΣΑΚ να μην είναι μόνο αφοσιωμένη, αλλά και ε, άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει αυτά τα θέματα εδώ και καιρό. Διαβίβασα στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου ε, την άποψη ότι θεωρώ ότι εσύ και εγώ θα πρέπει να προεδρεύουμε και σε αυτή την αντιπροσωπεία όπως και στην προηγούμενη και να μας συνοδεύσουν συνάδελφοι που παρακολουθούν το θέμα αυτό σε βάθος εδώ και καιρό και με κύρος. Και ένα τελευταίο σχόλιο που είναι επίσης ανισχυτικό, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να μας απασχολήσει πιστεύω. Αυτό που ε, καταλάβαμε στις συνεδριάσεις αυτές τι είναι. Θέλουν ο μηχανισμός ΚΟΖΑΚ να πριτανεύει όλων των σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίου. Ακόμα και για την παρακολούθηση αυτή την κοινοβουλευτική της Europol, της Eurojust, να είναι αυτός ο μηχανισμός. Από τη μια 162 και από την άλλη 6. Όχι, θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το μηχανισμό μια για πάντα και να πούμε ότι Είμαστε δύο ισότιμοι συνομιλητές και αυτή η ε, έννοια για μας είναι σαφής, για άλλους λιγότερο βέβαια. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία εμείς έχουμε μια μεγάλη δυσκολία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλούστατα, οι συνάδελφοί μας δεν πάνε στις συνεδριάσεις. Αν πιέζουμε εμείς να έχουμε 40% ή 33% συμμετοχή και τελικά φτάνουμε στις συνεδριάσεις και δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους συναδέλφους να πάνε. Όχι 30, ούτε 3. Ε, οπότε αυτομάτως, καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ασυνέπειας, να ε, το πω έτσι. Και δεν έχουμε εξασφαλισμένη παρουσία των συναδέλφων. Κάπως θα πρέπει να το δούμε αυτό. Οι πολιτικές ομάδες δεν ξέρω. Για να μην μας λένε, όπως μας το είπαν αυτό στη διάσκεψη των Πρόεδρων, ότι γιατί ζητάτε 33% αφού δεν πατάει ποτέ κανείς. Έτσι κι αλλιώς δεν έρχεστε. Τι το θέλετε το 33%. Αυτό δεν ισχύει στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές πάντα στις επιτροπές, αλλά στις συνεδριάσεις ε, τις διακοινοβουλευτικές σίγουρα συμβαίνει αυτό, γιατί οι συνάδελφοι έχουν και άλλες ενασχολήσεις και άλλες υποχρεώσεις και αυτό είναι εις βάρος ε, των κοινών μας ε, καθηκόντων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά ήθελα να σας πω και σας επαναλαμβάνω τις συμβουλές του Προέδρου ε, υπομονή, καρτερία ε, όχι βεβαιασμένες κινήσεις, αλλά δεν θα ήταν περιττό ή άσκοπο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για να δούμε πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την εμπλοκή, πώς να ανοίξουμε το δρόμο που είναι κλειστός αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση. Ε, ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας και για την καρτερία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρτίνε. Είμαι συγκινημένος και με εκπλήσουν όλες αυτές οι λεπτομέρειες που έμαθα, οι τόσο ιδιαίτερες, κυρίως ε, η διάμετρος ε, της μεγάλης ρόδας του βελοσιπέδου 162 εκατοστά ήταν το μικρό και η μεγάλη ρόδα και 6 η μικρή. Τέλο πάντων, υπομονή πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε μια ολόκληρη περιστροφή. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Γκουρμάη καταρχάς. Σα ευχαριστώ. πρόεδρε. Μόλι έμαθα ότι ε, η Εθνική, ε, το Εθνικό Κοινοβούλιο της ε, Ουγγαρίας ενέκρινε την μεταρρύθμιση του συντάγματος, υπερψηφίστηκε από το κυβερνητικό κόμμα, καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Έχουμε επομένως ένα νέο σύνταγμα στη χώρα μου και θα στο παρουσιάσει αύριο ο κύριος Σάιερ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό νωρίτερα όπως είχαμε ζητήσει άλλωστε. Ας επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή Ο συνήθως ο Μιχελάνκεφ Μαρτίνεθ θα είναι πάρα πολύ καλός στο να μας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στην ε, ΚΟΖΑΚ και γενικότερα για τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και Ξέρετε ότι από την προηγούμενη μα συνάντηση συνέβησαν πολύ ενδιαφέροντες εξελίξεις, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο στη στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια συζητήθηκε η σχέση που θα μπορούσε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια, καθώ και την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συζητήθηκε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την επιτήρηση του χώρου δικαιοσύνη και ασφάλειας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε, καθώς επίσης και η εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η επιτήρηση της Europol. Πέρα από αυτά όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και η επιπτώση που θα έχει στους εθνικούς προπολογισμούς. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε τα εθνικά κοινοβούλια και καταλαβαίνετε να φέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε στο ζήτημα αυτό καθώς επίσης και στο πολύ σημαντικό ζήτημα για διαφάνεια, το οποίο υπάρχει όλο και περισσότερο από του Ευρωπαίου πολίτε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο σημεία αφού διάβασα τα συμπεράσματα τη συνάντηση αυτή. Καταρχά, ε, υποστηρίζω πλήρω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνεια, καθώ επίση και κατάλληλη πληροφόρηση για του Ευρωπαίου πολίτε όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και πολλοί βρίσκονται σε πολύ επισφαλείς καταστάσεις λόγω της κρίσης. Πρέπει λοιπόν να τους δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της προκειμένου να ενδυναμώσει την οικονομική διακυβέρνηση και να προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Είμαι σαφώς υπέρ του να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα λιτότητας, μέτρα αυστηρότητας, αλλά και εκείνα τα οποία προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την έρευνα, προκειμένου να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικές κρίσεις, οι οποίες ε, θίγουν περισσότερο τους πιο ευάλωτους. Καταλαβαίνετε ότι η κρίση μας επηρεάζει όλους και μολονότι προχωρούμε όλοι τώρα σε μεταρρυθμίσεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανταπόκρισή μας στην κρίση θα πρέπει επίσης να βασίζεται και στην κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς επίσης σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Είμαι πεπισμένη ότι τα φόρα αυτά, όπως η κόζακ και η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας προσφέρουν τελικά τη δυνατότητα για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις στις υφιστάμενε αυτές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό ότι λάβαμε λοιπόν την ενημέρωση αυτή, ότι μπορέσαμε να σχολιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμω να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο προκειμένου να ενημερώσουμε και του πολίτες μας ότι πρέπει να καταφέρουμε να επιβιώσουμε μέσω της κρίσης. Ευχαριστούμε την κυρία Γκουρμάη. Ο κύριο Ντάφ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ για την εξαιρετική του δουλειά καθώς προασπίζεται τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Δεν είναι όμως θέμα προνομίων ε, και αρχών. Και εδώ έγινε και το πρόβλημα. Εάν δεν συμφωνήσουμε με μια νέα βελτιωμένη διαδικασία για τη διακυβουλευτική συνεργασία για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και την κοινή εξωτερική πολιτική, θα πληχθούν οι διαδικασίες. Και είναι σαφές ότι κάποια εθνικά κοινοβούλια αρνούνται ότι υπάρχει συνθήκη της Λισαβόνα και δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ε, αποτυχία και την ε, ε, πάυση της διαδικασίας των πυλώνων και δεν μπορούν να δουν ότι υπάρχει πλέον εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν κατάφορο σφάλμα από πλευράς μας να δείξουμε απλώς συγκατάβαση και να μην ε, αντιδράσουμε. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εκφράζουμε τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να κάνουν τα δικά τους καθήκοντα και δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη αυτή αποτελεσματικά. Επιπλέον είναι σημαντικό να σεβαστούμε τον δεταλμένο ρόλο των εθνικών κοινοβολίων στους τομείς αυτούς, αλλά το αντίτιμο είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει και τα ίδια με τη σειρά τους να αρχίσουν να σέβονται το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φρονώ λοιπόν ότι η προτινόμενη άγουσα, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του Προέδρου Μπούζεκ και του κυρίου Μαρτίνεθ, Μαρτίνεθ και της ομάδας εργασίας ε, για τη διακοινωνιοβουλευτική συνεργασία είναι η σωστή. Και δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα σε αυτό το στάδιο. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εξέφρασε την άποψή τους και στην έκθεση Αλμπερτίνη και στην έκθεση Γκουαλτιέρη. Δεν θυμάμαι βέβαια ποια από τις δύο ήταν αυτή που ε, ανέφερε μία παράγραφο η οποία αναφέρει ρητός ότι Λυπόμαστε που διεκόψαν οι συζητήσεις μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια το Μάιο θα ψηφίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις και θα περάσουν κατά πάσα πιθανότητα. Επομένω, θα έχει καταγραφεί και επισήμω η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ότι δεν συμφωνούμε με όσα συνέβησαν και θα παραμείνουμε εν αναμονή καλύτερων συνθήκων πριν ξεκινήσουμε εκ νέου πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και ημών. Αυτά νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ και εσείς ε, επισημαίνετε αυτή την πτυχή της καρτερίας που είναι αυτή που χαρακτηρίζει και τους ισχυρούς άλλωστε. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Μικελάν Χέλ Μαρτίνεθ, όχι τόσο για τις πληροφορίες που μας έδωσε σήμερα, αλλά και διότι μέσω αυτών των πληροφοριών μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πώς ε, είναι η κατάσταση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γεγονός ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις επαφές μας και να μην είναι τόσο απογοητευτικά τα πράγματα και ταυτοχρόνως ότι ε, προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Παρά το γεγονό ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση επικεντρώθηκε στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την ε, ε, πολιτική ασφάλεια και άμενα, θα ήθελα, επειδή δεν είμαι εμπειρογνώμων επί του θέματο, να επισημάνω κάτι το οποίο αναφέρατε κι εσείς, τη δύσκολη σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό απορρέει από κάτι το οποίο κανονικό θα έπρεπε να είναι θετικό στοιχείο, η αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία όμως από το 2009 κατέληξε να είναι επειδή εμείς ως ευρωβουλευτές δεν θεωρούμαστε εθνικοί βουλευτές, ε, παράγοντας ο οποίος μας απομάκρυνε διότι θεωρείται ότι κάνουμε κάτι εκδιαμέτρο διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή όπως έχει η ευρωπαϊκή κατάσταση ανθούν οι λαϊκισμοί οι οποίοι λαϊκισμοί είναι αντιευρωπαϊκοί. Το είδαμε αυτό, για παράδειγμα, στις φιλανδικές εκλογές, οι οποίες εξήχθησαν εχθές. Ε, το είδαμε και σε άλλες εκλογές, εκλογές αναμετρήσεις στην Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το διαπιστώσαμε και σε κάποιες ε, δηλώσεις ε, πολιτικών ηθινόντων από την Ιταλία, οι οποίοι έθεσαν ακόμα και θέμα εγκατάλειψης Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν επιληθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και εν δημιουργείται ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα το οποίο αποτελεί και τη βάση πολιτικών κινημάτων τα οποία λαμβάνουν και πολύ καλά ποσοστά σε εκλογές. Στην πράξη, στην πραγματικότητα, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βιώνουν οικονομικές περικοπές και κοινωνικά προβλήματα και πολλές φορές θεωρούν ότι οι πολιτικές ευρωπαϊκές σύνησες είναι υπεύθυνες για τις περικοπές και από την άλλη έχουμε χώρες οι οποίες είναι θύματα της καλής ζωής εντός εισαγωγικών ε, σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες πλήττουν την ευημερία των πιο προηγμένων χωρών. Θεωρώ ότι αυτό το κλίμα μεταξύ Ευρωπαίων εκπροσώπων αν θέλετε και εθνικών εκπροσώπων ε, δυστυχώς ε, δεν θα πρέπει να επιδεινωθεί και οι καλές σχέσεις είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη ρήξη που υπάρχει μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για να επανέλθω τώρα εντάχει στο θέμα της ε, εξωτερικής πολιτικής και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο ανταποκριθήκαμε στην κρίση στη Λιβύη εκφράζει με πολύ καλά ε, το πώς ε, ε, επειδή ακριβώ υπάρχει αυτή η σύγχυση και έχουμε χώρε που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, χώρε που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν στι δυνάμει που παρεμβαίνουν στη Λιβύη, αλλά μόνο με προστατευτικό τρόπο, άλλε είναι αυτέ που κάνουν την παρέμβαση. Υπάρχει λοιπόν μια πολύπλοκη κατάσταση και δυνητικά μπορεί να αρχίσουν ε, να υπάρχουν διαρροές και να μην υπάρχει πολιτική συνένεση και να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και όπως επεσήμενε ο Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να είναι μόνο η Κόζακ. θα πρέπει να έχουμε ένα ad hoc ε, ε, εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέπει να τη δράσουμε. Ολοκληρώνοντας να πω ότι θα πρέπει πράγματι να μάθουμε να χορεύουμε από κοινού, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να χορεύουμε και γρήγορα και με συνέπεια. Και αυτό σας το λέω διότι αν χρησιμοποιήσουμε μόνο την καρτερία και τη σοφροσύνη, μάλλον θα προσεγγίζω πιο πολύ τι απόψει του ΕΛΚ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λέω συνέπεια ε, για να καλύψουμε και τις υπόλοιπε ομάδε ε, ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Και η συνέπεια όμως είναι κόρη της καρτερίας. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ και εγώ τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες Μαρτίνες για την έξοχη δουλειά του και για την ε, καλή συνεργασία που είχε με την περιορισμένη αυτή ομάδα η οποία ανέλαβε να καθορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου επί του θέματος. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στην επόμενη ΚΟΖΑΚ. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πολύ σαφή στοιχεία αυτή τη στιγμή και σε κάποια από τα στοιχεία στα οποία στην ε, διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων ε, καταλήξαμε σε συμφωνία, τα οποία είναι σημαντικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι συμφωνούν ότι η διάσκεψη αυτή όταν θα συσταθεί δεν θα εκπώνει γνωμοδοτήσεις, αλλά απλώς ε, θα καταλήγει σε συμπεράσματα μέσω συνένεσης, προκύπτει σαφώς ότι έγινε κατανοητό ότι δεν υπάρχει κενό κοινοβουλευτικού ελέγχου το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε με νέο όργανο, αλλά υπάρχει ανάγκη για συζήτηση, συντονισμό και αντιπαράθεση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο καθένας ασκεί ένα τμήμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως δεν υπάρχει ένα νέο όργανο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει ένα κενό, αλλά υπάρχει συντονισμός μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο καθένας με τη σειρά του στη συνέχεια ασκεί το θεσμικό του ρόλο στο επίπεδό του, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα Εθνικά Κοινοβούλια σε, εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, τα, εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν ε, αντιληφθεί σαφώς το ρόλο τους, παρόλο που θέλησαν να το συμπεριλάβουν στο τελικό έγγραφο. Δηλαδή, εάν δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα νέο όργανο, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα χώρο συζήτηση και αντιπαράθεση, θα πρέπει αυτό ο χώρο να καθοριστεί βάσει των ε, αντίστοιχων προτεραιοτήτων που είναι εντέ και για την περίπτωση των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτό είναι προφανέ, αλλά και για την ε, περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ο προπολογισμό, η υπατή εκπρόσωπο, οι αποστολέ, οι οποίε συνήθω είναι πολιτικέ αποστολέ, κυρίω όσον αφορά τι αμυντικέ δαπάνε, το Κοινοβούλιο χρηματοδοτεί ένα μικρό ποσοστό, το διοικητικό κόστο ε, σε επίπεδο Βρυξελών ε, για τι στρατιωτικέ δαπάνε, για την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Πρόκειται λοιπόν για αρμοδιότητες οι οποίες είναι σημαντικές εκατόρθεν αλλά και ε, όσον αφορά και το συνταγματικό του ρόλο όπω καθορίζεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Όπω θα σα πει και ο κύριο Ντάφ σε λίγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται ω το όργανο στο οποίο υπάρχει άμεση εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι λοιπόν ένα εθνικό κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους ε, πολίτες της κάθε χώρας συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει ο άμεσος και ο εθνικός τρόπος εκπροσώπησης. Θεωρητικώς λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε 50 και 50 εκπροσώπους, αλλά επειδή εμείς συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ανάγκη να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, δεχτήκαμε να είμαστε κάτω από το 50-50 και μάλιστα ουσιαστικά κάτω. Αλλά βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και ένα κατώτατο όριο. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να μιλάμε για ποσοστά και όχι για απόλυτους αριθμούς και θα πρέπει να παραμείνουμε στην πρόταση του ενός τρίτου και να φτάσουμε ίσως ως χείριστη περίπτωση στο 20% εάν θέλουμε οπωσδήποτε να καταλήξουμε στο συμβιβασμό. Οτιδήποτε κάτω από το 20% θα ήταν αδύνατο για μας. Το 20% ούτως ή άλλως είναι το ίδιο ποσοστό εκπροσώπηση που έχει το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Επομένως είναι ουσιαστικό σημείο αναφοράς. Δύο θέματα για να ενισχύσω αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Ματίνης, Η καρτερία, το είπαμε αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πολύ σταθεροί για να έχουμε ένα πρώτο πρωτόκολλο Το άρθρο 10 έρχεται μετά από το άρθρο 9. Επομένως, οτιδήποτε έχουμε θα πρέπει να καθοριστεί μέσω συνένεσης, κοινή συμφωνίας. Εάν λοιπόν αποφασίσουν κάτι μονομερό στα εθνικά κοινοβούλια, αντιβαίνουν στη συνθήκη. Και επ' αυτού εμείς θα πρέπει αφενός να επαναλάβουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε ε, ε, από κοινού αυτή τη διάσκεψη και επίσης να διευκρινίσουμε ότι το άρθρο 9 λέει σαφώς ότι οποιαδήποτε μορφή τακτικής συνεργασίας θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων και δεν καθορίζεται μονομερός. Συμφωνώ λοιπόν ότι για αυτές τις αρχές υπάρχει ευρύτερη συνένεση στο Κοινοβούλιο. Αυτά που μας είπε ο Πρόεδρος Μαρτίνες αντικατοπτρίζουν την άποψη των βασικών πολιτικών ομάδων. Επομένω αυτό που μας προτείνει ως ε, οδό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκουαλτιέρη. Ο κύριο Σέπφλιν. Uh, σα ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα όντω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ Ε, μου προκαλεί εντύπωση αυτή η μεταφορά που χρησιμοποιήσατε για τον χώρο, γιατί αυτό το οποίο δεν αναφέρατε ήταν ότι ε, υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στο χορό. Κάποιοι οποίοι θα μένουν εκτός του χορού τόσοι ή άλλως. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Μου έκανε εντύπωση επίση η ε, εισαγωγή, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική. Αναφερθήκατε όντω στην υφιστάμενη κατάσταση αδιεξόδου. Υπάρχει έντονη τριβή, πολλέ εντάσει είπατε και θα μπορούσα να θέσω πολλέ ερωτήσει ω προ αυτό η ε, εχθρότητα αυτή, το επίπεδο αυτό ε, εχθρότητα στο οποίο είδατε είναι δική σας προσωπική εκτίμηση, είναι κάτι το οποίο υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενδεχομένως να έφτασε σε ένα νέο κρεσέντο αυτή τη στιγμή. Αποτελεί απόρρια τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, μέσω της οποίας τα εθνικά κοινοβόλια συνειδητοποιούν πλέον περισσότερο ότι όντως υπάρχει μια ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι δεν απαραίτητα ικανοποιημένα με την κατανομή αυτή. Επίσης, περιορίζεται αυτό μόνο στο πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε, δηλαδή τη κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ή έχει να κάνει με κάτι βαθύτερο και ευρύτερο. Γιατί μόνο, αν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τότε καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχει μία διάσταση τόσο ευρωπαϊκή όσο και εθνική. Και οι δύο είναι νόμιμες και οι δύο είναι κέρυες. Βέβαια, χωρίς την ευρωπαϊκή διάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά ο μηχανισμός, γιατί ε, το ίμιση των προτάσεων, το ίμιση του μηχανισμού ουσιαστικά θα απουσιάζει. Αν λοιπόν υποβάλουμε το επιχείρημα αυτό ότι χρειαζόμαστε μεν του δε, αν καταφέρουμε να προωθήσουμε το μήνυμα αυτό, το νομίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή πλατφόρμα βάσει τη οποία θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστούμε. Κύριε Σέπφιλ, κοιτάξτε, εμείς εδώ δεν αναφερόμαστε εν γέννη για την οικονομή, στην οικονομία και σε προβλήματα ισονοσημασίας. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνα. Είναι το βασικό στοιχείο που αποτελεί την ενότητά μας. Ή έχουμε ενότητα ή δεν έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι η ιδέα μιας κοινή ε, άμυνας ήταν αυτή η οποία έδωσε την αίθουση για την Ευρώπη και αυτή η επιμονή μας μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όμως αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Μαρτίνες για την παρουσίαση των προβλημάτων. Πολύ ειλικρινής ήταν και ανοιχτός ο λόγος του. Νομίζω θα πρέπει να ψάξουμε όμως ακόμα πιο βαθιά τα αίτια. Γιατί δεν είναι μόνο η ουσία, είναι και ο τύπος εδώ της συνεργασίας. Και αν θέλετε να παραμείνουμε σε αυτή τη μεταφορά, μπορεί να χορεύουν δύο παρτενέρ μεταξύ τους, αλλά ο ένας πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και ο άλλος προς την άλλη. Και πού να βρεις ρυθμό εκεί. Και δεν καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και το ρυθμό, αλλά και τη μουσική. Και αυτό να συζητήσουμε και την ουσία του θέμα ε, θέματος της συνεργασίας Εθνικών Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι εγώ πιστεύω και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ για την εξωτερική πολιτική και την ΚΕΠΑ. Ε, θα το δούμε και αλλού αυτό. Και με ανησυχεί ω τάση αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε μήπως καμιά φορά φταίμε και εμείς για τον ε, τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι στην Ευρώπη. Όταν συζητήσαμε για το Europlus, αυτό το σύμφωνο για το ευρώ, που συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα πριν ζητήσουμε συνεννόηση με τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες για να βολιδοσκοπήσουμε και να δούμε ε, οι απαντήσεις που τους προτείνουμε ανταποκρίνονται ε, στις ανησυχίες, τα μελήματα, τα προβλήματά τους. Αυτό εμένα με βασανίζει. Η κοινοτική μέθοδος, την οποία εμείς πρεσβεύουμε εδώ και εκπροσωπούμε βρίσκει αποδοχή στα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και των κυβερνήσεων των κρατών μελών και ε, της ευρεία δημόσιας συζήτησης που γίνεται στις χώρες. Καλή υπομονή, αλλά να δείξουμε και μια ανυπομονησία ως προς τον τρόπο με τον οποίο εμείς προβάλλουμε τα ευρωπαϊκά θέματα στους Ευρωπαίους πολίτες, στην κοινή γνώμη και πώς εκείνοι τα αντιλαμβάνονται. Και για την ΚΕΠΑ, ακριβώς είναι περίπλοκη εκεί η συνεργασία, η κοινοβουλευτική, μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι και ενδεικτικό αυτό για τη διχόνοια που μας μαστίζει και τα ημίμετρα που παίρνουμε. Γιατί τελικά ε, καταλαβαίνουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θέλει να εκχωρήσει εξουσίες και αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σε αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει κοινοτικοποίηση. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να συναντηθούμε και με τα κοινοβούλια για το ποιο τα ελέγχει αυτά τα θέματα. Και για να μην ρίξουμε νερό στο μήλο των λαϊκιστών, θα πρέπει να συζητάμε και το περιεχόμενο και την ουσία για το τι συναποφασίζουμε, αλλά να συζητούμε και τα άλλα θέματα και τον τύπο της συνεργασίας. Θα πρέπει ο τύπος να συναντάει την ουσία για να προχωρήσουμε αποτελεσματικά στη συνεργασία μας και στην ΚΟΖΑΚ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια. Και τέλος, να πω και το εξής οποιαδήποτε αναζήτηση δημιουργίας μιας τρίτης δομής, κοινοβουλευτική συνέλευση που θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ασφαλείας, το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Γιατί θολώνει ακόμα περισσότερο τα νερά και τη δουλειά και του Εθνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το σταματήσουμε αυτό το εγχείρημα, το κόψουμε εδώ. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, στη συνάντηση των Βρυξελών δεν περάσατε σε πολύ ουσιώδη ζητήματα, αλλά ασχοληθήκατε κυρίως με διαδικαστικά ζητήματα. Και αν κατάλαβα καλά, Φαίνεται ότι ε, ένα σημείο επί το οποίο υπάρχει συμφωνία είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μειώσει την εκπροσώπησή του από το 14% στο 4% αν δεν κάνω λάθος. Επομένως το μήνυμα για μένα είναι ξεκάθαρο είτε θέλουμε το δεχτούμε είτε όχι, ότι ε, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των ε, εθνικών κρατών μελών πιστεύουν ε, ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια δεν αποτελεί νόμιμη αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ακόμα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνάδει ούτε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ούτε με προηγούμενε συνθήκε. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε και ακόμα στο Μάστριχτ. Από ό,τι φαίνεται όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο ή άδειλα επίση και οι ίδιε οι κυβερνήσεις. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν το μήνυμα αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πολλοί ε, ομιλητέ αναφέρθηκαν σε λαϊκισμό, σε λαϊκιστικέ στάσει, με ιδιαίτερη γραφικότητα και από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιούν το επιχείρημα αυτό όλο και περισσότερο κάθε φορά που αναφέρονται στη δημοκρατία. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο πολλές φορές δημοκρατικά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ως λαϊκίστικα, όπως για παράδειγμα το πρώτο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία χαρακτηρίστηκε λαϊκίστικο, το δεύτερο βέβαια αποτέλεσμα δημοκρατικό. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, και τώρα ο συνάδελφος Μαρτίνης για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα πράγματα μπορώ να πατήσω συγκεκριμένα και άλλα γενικότερα. Στον κύριο Μπρόνς πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, ε, έχετε δίκιο κύριε Μπρόνς όταν λέτε ότι ε, είναι αλήθεια στα θέματα ασφάλειας και άμυνας από πολλούς εκφράστηκε η άποψη ότι αυτά δεν είναι αρμοδιότητα, ούτε πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός αυτό ότι υπόθηκε. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτοί που έλεγαν αυτά τα πράγματα πολύ εύκολα θα σας πούνε ότι τίποτα δεν χρειάζεται να είναι ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρνούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ύπαρξή του την ίδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια, φυσικά θα σας πούνε ότι ούτε στην ΚΕΠΑ έχουμε αρμοδιότητα αφού δεν θέλουν την Ένωση. Και ότι τι ανακατεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τη πέφτει λόγο. Και ε, αρχίζει γενομένης από την ΚΕΠΑ πάνε και πιο πέρα. Και σε άλλους τομεί πολιτική σιγά σιγά επεκτείνονται. Αυτή είναι η θέση τους. Δεν λέω ότι είναι αθέμητη η άποψη. Δυστυχώ όμω όλο και περισσότερο γενικεύεται σε πολιτικούς τομείς και χώρους που αποκτούν σημασία στις χώρες μας. Άλλο είναι βέβαια ότι εγώ ε, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, ενώ ορισμένοι άλλοι χαίρονται. Επίσης, κάποιοι συνάδελφοι είπαν, και σωστά, ότι αυτό το πρόβλημα διαφωνίας ή διάστασης ε, απόστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα Εθνικά Κοινοβούλια αντανακλά το κύμα επανεθνικοποίησης που σαρώνει τώρα την Ευρώπη. Η απόρριψη της κοινοτικής μεθόδου και οι προσδοκίες ορισμένων που ακόμα δηλώνουν βέβαια ευρωπαϊστές. Οι ευρωπαϊστές έτσι, όχι οι αντίπαλοι της Ευρώπης, αλλά πολλοί από τους οπαδούς της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό που χρειάζεται για να χτιστεί η Ευρώπη είναι ένα συντονισμός και μάλιστα διακυβερνητικός, χωρίς να το πάμε παραπέρα. Και βέβαια σε αυτό το οικοδόμημα δεν υπάρχει ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να γυρίσουμε πίσω 50 χρόνια, να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα είναι ένα συντονιστικό όργανο, λέει, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό το όραμα μπορεί να είναι θεμητό, αλλά δεν είναι το δικό μου, εν πάση περιπτώσει. Και είναι ένα όρεμα ανιστόρητο τουλάχιστον να το αναγνωρίσουμε. Και κάθε φορά, είτε μας αρέσει είτε ε, όχι, γνωρίζει όλο και περισσότερο ε, υποστήριξη. Είτε είναι λαϊκισμός είτε δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η Βρετανία, ας πούμε, εκπρόσωποι και της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων και οι αντίστοιχοι πρόεδροι κάποια στιγμή συζητούσαμε μαζί τους για μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Και έκαναν λάθος και τις δύο φορές είπαν διακυβερνητική διάσκεψη. Και τους είπα σας πρόδωσε ο Φρόιντ αγαπητοί συνάδελφοι. Λανθάνουσα γλώσσα αλλά το είπανε. Διακυβερνητισμό θέλουν. Δεν λέω ότι είναι αθέμητο. Λέω ότι δεν το θέλω εγώ και, για μένα είναι οπισθοδρόμηση ε, στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση τα τελευταία χρόνια. Και ανησυχώ έτσι με κάποια έννοια. Γιατί ορισμένοι μυθοποιούν ε, την ε, συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης τη Μακαρίτησα. Και τη μυθοποιούν γενικά. Αυτοί που τη μυθοποιούν δεν τη γνωρίζουν. Εγώ διατέλεσα επί δεκαετία αντιπρόεδρο τη συνέλευση αυτή και ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο ήταν ο ρόλο κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκούσαμε αυστηρού κτλ. Σιγά μην κάναμε κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ποτέ στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση έτσι, με αυστηρό τρόπο. Και όποιο θα υποστηρίζει αυτά, ε, είτε κοροϊδεύει τον εαυτό του, είτε δεν ξέρει περί τίνο ε, μιλεί. Δεν λέω ότι δεν ήταν ενδιαφέρον το θεσμικό όργανο. Εντάξει, αλλιώς δεν θα άντεχα κι εγώ 20 χρόνια μέλος και 10 χρόνια αντιπρόεδρος. Και είναι και εδώ ορισμένοι παρόντες που τα ξέρουν και είχε και καλούς υπαλλήλους, εντάξει. Αλλά δεν είναι ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος αυτό που κάναμε. Ποτέ δεν ήταν. Και το έχω ξαναπεί και το έχω πει και στους φίλους τους Βρετανούς. Ούτε μία φορά δεν υπήρξε ψήφισμα της ε, ΔΕ, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, που να είχε συζητηθεί στα εθνικά κοινοβούλια. Σε καμία βουλή σε κανένα σώμα Εθνικού Κοινοβουλίου. Εγώ το προσπάθησα στη Βουλή της χώρας μου γιατί θεώρησα ότι ορισμένα ψηφίσματα μπορεί να ήταν ενδιαφέροντα για τους βουλευτές. Ε, εντάξει όμως, ας μην ε, υπερβάλλουμε. Κοιτάξτε, ποια είναι τα δύο πιθανά σενάρια που θεωρώ εγώ ότι διαγράφονται. Και το έχω ξαναπεί και το λέω χωρίς καμία επιθετικότητα. Σας είπα, το πρώτο σενάριο να είναι ένα ποδήλατο ασύμετρο από τα παλιά ποδήλατα του 19ου αιώνα ή θα είναι ένα σύστημα ισότιμο που θα στέκει στα πόδια του, ο ένας θα εμπλουτίζει τον άλλον, θα συνεργαζόμαστε και πάλι ε, από το ρόλο το διακριτό του καθενός, τον ξεχωριστό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει κοινοβουλευτικά ή παρακολουθεί εν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο και παρακολουθούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους. Εάν θέλετε, εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί θα πρέπει να βρούμε τη σύνδεση, να αγκιστρωθούμε. Και βέβαια έχει δίκιο ο κύριος όταν λέγει ότι θα πρέπει να διδαχθούμε Βεβαίω και για το χορό που σα είπα, μαθαίνει κανεί να χορεύει. Και μαθαίνει να σέβεται και τον παρτενέρ. Δεν θα το τραβά από το λαιμό, ούτε θα το καταπατά, ούτε θα τον σέρνει. Ο χορό σημαίνει αρμονία και σεβασμό. Και εγώ πάντα σέβομαι και προσπαθώ να σέβομαι την παρτενέρ μου, με την οποία χορεύω. Ο κύριος Μέντε δεν φύγω με αμφισβητεί και με εκπλήσει. Ε, για ποιο λόγο, πώς σας ήρθε αυτό. Λοιπόν, ο συνάδελφος και φίλος Εύλιν ρώτησε κάτι και νομίζω ότι λίγο απαντήσαμε σε αυτό ήδη. Σε γενικές γραμμές επικρετεί ένταση. Ή ε, πώς να το πω. Επιφυλακτικότητα με σκεπτικισμό βλέπουν τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα αυξανόμενο, προφανέστατα. Και γίνεται και πιο οξύ σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί εμάς, βεβαίως, της ασφάλειας, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Διότι είναι γεγονός ότι αυτοί οι τομείς ε, κατεξοχήν είναι αρμοδιότητα εθνική και υπόθεση των κρατών και των κοινοβουλίων τους. αλλά είναι προφανές ότι αυτό επεκτείνεται περισσότερο. Είναι κάτι, έτσι, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και υποβόσκει το ρεύμα επανεθνικοποίησης, διακυβερνητικής συνεργασίας, άρνησης ε, της κοινοτικής μεθόδου που το είπαν για κάποιοι συνάδελφοι. Και τελειώνω λέγοντας κάτι που είπαμε και προηγουμένως. Δύο είναι τα σενάρια. είτε θα είναι τα δύο σώματα που θα συνεδριάζουν και θα συνεργάζονται με τρόπο αρμονικό, με σεβασμό, και το άλλο σενάριο είναι το εξή. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, όπως κάνουμε μέχρι τώρα, στην Επιτροπή Εξωτερικών, στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, ε, στην άλλη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά. Και τα Εθνικά Κοινοβούλια, από την πλευρά τους, θα ορίσουν, θα φτιάξουν ένα συντονιστικό όργανο, χωρίς εμείς να συμμετέχουμε καθόλου, που να εργάζεται, να λειτουργεί και αυτό το συντονιστικό τους όργανο θα αποφασίζει αν θα συνεδριάζει δις ή δεκάκι, ξέρω εγώ, ή αν θα έχει δύο γλώσσες ή δέκα γλώσσες, ή αν θα έχουν 50 προσώπους ο καθένας ή δύο, χωρίς εμείς να έχουμε καμία ανάμιξη. Και αν μας καλέσουν ως παρατηρητές, θα πάμε παρατηρητές. Αυτά είναι τα δύο πιθανά σενάρια. Δεν υπάρχει άλλο. δεν βλέπω. Τι συμβαίνει. Σε αυτή την προοπτική θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ σε μια επιτροπή σαν τη δική σας και στους παρόντες συναδέλφους ότι μέχρι τώρα και στο σενάριο Κοζάκ κατά κύριο λόγο με μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόμασταν με έναν τρόπο που νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το πάμε έτσι. Στην ΚΟΣΑΚ εμεί είμαστε μέλη, είμαστε αναπόσπαστο τμήμα, αλλά είμαστε ένας από 28, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι κάνουμε συνεδριάσεις όπου οι άλλοι 27 εταίροι, ας πούμε, παράγουν κάτι δηλώσεις ή έγγραφα επιθετικά και εχθρικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, όσο καλόπιστος και να είσαι, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και αξιέπαινη ε, των υπαλλήλων μας και των συναδέλφων μας και ημών, προχωρήσαμε και μπορεί στην αρχή ε, να ήταν οξύτατη η κριτική και σφοδρότατη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταφέραμε το 95% να φύγει της κριτικής και να παραμείνει το 5% και τελικά το υπογράψαμε το έγγραφο. Από εδώ και στο εξή εγώ σας λέω ότι σε, ό,τι με αφορά δεν παίζω πια, δεν μπορώ να δέχομαι και να καταπίνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπογράφει ένα χαρτί που κατά 5% επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ένα σώμα εθνικών κοινοβουλίων να βγάζει ένα χαρτί πάρα πολύ εχθρικό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα απαντήσει. Αλλά όχι να υπογράφει και το Κοινοβούλιο την κριτική. Όσο μετριοπαθής και να είναι, ως προς το τι εστί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το τι πράττει. Δεν μπορεί να το υπογράφει. Εγώ δεν το προσυπογράφω πια και, δεν είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και νομίζω και ο κύριος Κασίνη και οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε αυτά. Ούτε να λέμε ότι εντάξει, περιορίσαμε το έγγραφο στο 5% γιατί ήταν υβριστικό κατά 100% και τώρα δεν είναι υβριστικό, απλώς υπενήσεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρω εγώ, προσπαθεί να παρακάμψει ή να υπονομεύσει τις διακυβερνητικές σχέσεις. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος στο εξή μέσα στην ΚΟΣΑΚ να δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Να υπογράφει το Κοινοβούλιο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις δικές μας ψήφους αυτά τα πράγματα. Μάλλον έχουν παρεξηγήσει την καλή μας θέληση και τον τρόπο συνεργασίας και λειτουργίας που θέλουμε. Κάποιος είπε, νομίζω ο κύριος Νταφ, που πάντα είναι άκρος ε, ακριβής και μέγας οραματιστής. Είπε λοιπόν ότι είναι σαφές αυτόν τον καιρό ότι τα εθνικά κοινοβούλια βιώνουν περίεργες στιγμές δεν έχουν χωνέψει τη συνθήκη. Δεν έχουν κάνει κτήμα τους τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ή δεν το κατάλαβαν ή δεν συμφωνούν. Πάντως δεν το έχουν εστερνιστεί το κείμενο. Γιατί εμείς τι ζητούμε εδώ. Ούτε τίποτα παραπάνω, ούτε τίποτα λιγότερο ε, από εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Όχι με την σφιχτή έννοια, με την απόλυτη έννοια, με λογικούς μηχανισμούς. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουν χωνέψει τα κοινοβούλια, έχουν αυτό το ρεύμα της επανεθνικοποίησης, της διακυβερνητικής συνεργασίας, πράγμα όμως που είναι σύμβατο με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σας. Όταν έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας, <laughs> ζηλεύω που δεν είμαι μέλος. Τι να κάνω δεν μπορεί κανείς ε, ε, να είναι απανταχού παρά... Ξέρετε ότι στα γαλλικά υπάρχει παροιμία ότι δεν μπορεί να είσαι και στο μήλο και στο φούρνο. Να κάνεις και το αλεύρι και τα γλυκά. Ε, πάντως παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις ε, και από αλλού ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να σας αφουγραζόμαστε και σας είπα και στην αρχή ότι θέλουμε να μας προσανατολίζετε, να μας δίνετε ιδέες, γιατί ιδέες χρειαζόμαστε και έμπνευση, όχι μόνο υποστήριξη στα λόγια, αλλά καθημερινή στήριξη σε μια πολιτική που θα είναι δύσκολη η φάση. Α, συγγνώμη, Κάρλο. Κάποιος είπε ότι ένας μηχανισμός για να βρούμε λύσεις είναι να δουλέψουν περισσότερο οι πολιτικέ ομάδε, οι πολιτικέ οικογένειε. Το είπε και ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικέ παρατάξει ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ομοειδεάτε του στα εθνικά κοινοβούλια. Εντάξει, δεν χωράει καμία αφιβολία ότι και αυτή μια ιδέα είναι στα χαρτιά ωραία. Αλλά επειδή εδώ είμαστε πολύ παλιέ καραβάνε και τα ξέρουμε, φοβάμαι ότι θα είναι περιορισμένη η επιτυχία ίσως θα πρέπει πάντα να σκεπτόμαστε ότι τις, ε, οι εντάσεις οφείλονται σε διαφορά αντίληψη, σε διαφορά συμπεριφοράς. Εντάξει, δεν ξέρω. Εμείς φροντίζουμε ε, αυτό τον καιρό να είμαστε προσεκτικοί, καρτερικοί, χωρίς καμία υπεροψία. Ε, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε όλα. Υπήρξαν εθνικά κοινοβούλια που όταν είπαμε και πού θα συνεδριάζει αυτό το πράγμα, οπουδήποτε εκτό Βρυξελών και αν είναι στη Βρυξέλλε, οπουδήποτε εκτό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πάμε και στο Συμβούλιο να συνεδριάσουμε. Τίποτα άλλο θα μας πούνε. Ωραία ανέκδοτα. Ξέρω εγώ, μαύρο χιούμορ. Άλλοι είναι πιο πονηροί. Λένε, όχι, να συνεδριάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διερμηνία των καφέ και το πουρο όχι γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα, τι να κάνουμε. Ε, είναι πολύ διατεθειμένοι να συνεδριάζονται εδώ όταν εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ε, και αυτό το αστείακι θα πρέπει να σταματήσει. Ούτε λογικό είναι, ούτε μπορούμε εμείς πάντα να υπομιζόμαστε όλο το κόστος. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Μαρτίνεθ. Η κυρία Γιαννάκου ήθελε το λόγο. Λίγο σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Αντιπρόεδρος κύριος Μαρτίνες, ο οποίος έχει θητεύσει βέβαια στο Εθνικό Κοινοβούλιο, ε, είπε αυτό πραγματικά συμβαίνει. Ε, και εγώ επειδή έχω κάνει τέσσερις θητείες στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε διάφορα άλλα όργανα, νομίζω ότι πρώτον η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει καταργηθεί από πολλού χρόνου. Δεν έχει κανένα νόημα, παρέμενε μόνο για να γίνονται ταξίδια από τους εθνικούς βουλευτές. Και ιδιαίτερα από ορισμένε ομάδες που ήταν μόνιμες σε πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερον, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν όλες τις προβλέψεις μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας για να μπορούν να παρεμβαίνουν σε θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή πολιτική εγώ σας προτείνω να μην αναμειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε αυτή την υπόθεση. Να αφήσει τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν έναν συντονισμό όπως θέλουν να έχουν και αν και όταν χρειάζεται να υπάρχει επικοινωνία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είτε της Υποεπιτροπής για την Άμυνα και την Ασφάλεια ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλιώς θα είναι πάλι μια ατέλειωτη συζήτηση ε, χωρίς αποτέλεσμα, με συγκρούσεις, διότι κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα στις μεγάλες χώρες, οι εθνικοί βουλευτές δεν θέλουν ούτε να ακούνε για ευρωβουλευτές. Στις μικρές χώρες πρέπει να σας πω δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Είναι πιο καλό το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά εγώ προσωπικά έχω παραστεί σε συναντήσεις ε, Βρετανών συναδέλφων του Εθνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόκειτο για τον πόλεμο των μυρίων. δηλαδή υπάρχουν σημαντικές συγκρούσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναμειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει όλα τα όργανα που του διατίθενται για να κάνει τη δουλειά του και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και αν χρειάζονται συμπληρωματική συνεργασία αυτή μπορεί να γίνει. Αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας έχουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στα εθνικά κοινοβούλια, υπάρχουν Υπουργοί Άμυνας, υπάρχουν Υπουργοί Εξωτερικών. Εμείς δεν έχουμε απόλυτη αρμοδιότητα παρέμβασης, έχουμε όμως πολιτική αρμοδιότητα και πολιτικό βάρος και νομίζω να κάνει ο καθένας τη δουλειά του χωρίς να εμπλακούμε και πάλι με ένα καινούριο όργανο το οποίο μόνο σχόλια στην εποχή μας θα επισύρει για καινούρια έξοδα και για ταξίδια. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Νομίζω πάντως ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη συζήτηση λήξασα. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Εγώ κρατώ ε, το αριθμητικό στοιχείο από τα όσα μας είπε ο κύριος Μαρτίνες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το να θέλει κάποιος να πετάξει, αν θέλουμε να συντονιστούμε, και εδώ θα πρέπει να πω ότι το πρώτο πρωτόκολλο μας ζητάει να υπάρξει διακοινοβουλευτικό συντονισμός κυρίως διαρθρωμένο στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ. Θα πρέπει όμως ο συντονισμός να εκφράζει και μια ενιαίο προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένο αριθμό. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα όσα μας είπε ο κ. Μαρτίνα, παρά το γεγονός ότι σήμερα, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να έχει αίσιο τέλος στη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Πρέπει να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο πρόταση τροποποίησης ε, της πράξης της 20 Σεπτεμβρίου του 1976 για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία. Την ε, περασμένη Πέμπτη στο Στρασβούργο ακούσαμε τον ε, κύριο Νταφ ε, που έκανε συγκεκριμένε προτάσει συμβιβασμού και η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή. Ο εισηγητή τώρα μα έχει με ένα κατάλογο ψηφοφορία με κάποιε τροποποίησει, νομίζω κάποιε ή και προφορικό για τις συμβιβαστικές τροποποίησεις Επομένω επομένως του δίνω τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντά. κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες ήρθαν σε επαφή μαζί μου ζητώντας μου αν είναι απαραίτητο να ψηφίσουμε στην ε, Ολομέλεια του Μαΐου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να ζητήσουμε μία παράταση μέχρι τον Ιούνιο για να ψηφίσουμε δηλαδή στην ε, Ολομέλεια τότε. Νομίζω ότι ε, πρώτα βέβαια θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή, άλλωστε ψηφίζουμε αύριο, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι θα διακόψουμε στη συνέχεια για το Πάσχα, μετά έχουμε μια πράσινη εβδομάδα και καταλαβαίνετε ότι το όλο πακέτο μέτρων είναι πολύπλοκο και ιδιαίτερα μεγάλο, πιστεύω ότι θα ήταν πιο λογικό, πιο φρόνιμο να ζητήσουμε μια παράνταση και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου. και νομίζω ότι και οι σκιώδη εισηγητέ και οι συντονιστέ όλων των άλλων πολιτικών ομάδων συμφωνούν με την πρόταση αυτή. Δεύτερον, θα ήθελα γρήγορα να επιβεβαιώσω το ότι κατάφερα να βελτιώσω τις συμβαστικές τροπολογίες που συζητήσαμε στο Στρασβούργο στις 7 Απριλίου. Η συμβαστική τροπολογία Β δεν αναφέρει πλέον την αναφορά στον συνολικό αριθμό του μόνιμου πληθυσμού, η συμβαστική τροπολογία L LJV δεν αναφέρει πλέον την αναφορά στο σύστημα προτιμησιακής ψήφου με ήμια ανοιχτή λίστα. Επομένως, το όλο ζήτημα μεταξύ κλειστών καταλόγων και ή ανοιχτών καταλόγων παραμένει ανοιχτό για μια περαιτέρω διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Τρίτον, μετά από αίτημα του κυρίου Γκουαλτιέρη για το άρθρο 6 της πράξης, θα ήθελα να διατηρήσουμε την υφιστάμενη πρώτη παράγραφο, η οποία αναφέρεται στα μέλη του Κοινοβουλίου που ψηφίζουν σε ξεχωριστή και ατομική βάση. Αντί λοιπόν να αντικαταστήσουμε την πρώτη αυτή παράγραφο, τη συμπληρώνουμε τώρα με μία τροπολογία, την υπαριθμόν 7, την οποία έχω υποβάλει. Τέταρτον, όσον αφορά το ζήτημα των μειονοτήτων, θα έχουμε την ε, ευκαιρία να ψηφίσουμε για όλους τους επιθετικούς προσδιορισμούς, δηλαδή γλωσσικές και εθνοτικές μειονότητες, καθότι προβλέπεται εδώ πέρα ένα τρίτο ξεχωριστό τμήμα όσον αφορά την ε, ρήτρα αυτή, που αναφέρεται στην νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Και τέλος, συμβαστική τροπολογία J, J, ο κύριος Γκουαλτιέρη μου ζήτησε να αφαιρεθεί η διάταξη αυτή η οποία αναφέρεται στην ε, εφιστάμενη σύνθεση του Κοινοβουλίου καθότι δεν συνάδει η σύνθεση αυτή με την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Εγώ εξέφρασα βέβαια την προτίμησή μου να διατηρήσουμε την φράση αυτή στο κείμενο. Θα έχετε πάντως την δυνατότητα να διαφωνήσετε μαζί μου εφόσον τοποθετηθείτε διαφορετικά. Προσπάθησα να καταλήξω σε κάποιες σημαντικές συμβαστικές τροπολογίες μέσω της σύνταξης και επανασύνταξης της έκθεσης αυτής. Καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολο για ορισμένους από εσά να παρακολουθήσετε όλες τις διαδοχικές αλλαγές που συνέβαιναν στο κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υπομονή που έδειξαν, καθότι βλέπετε ότι καταφέραμε σιγά σιγά να καταλήξουμε σε μία τελική συνταγή για αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο προτείνουμε. Είναι σημαντικό στην παρούσα φάση να συνεχίσουμε να βλέπουμε τη σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Ακόμα θα υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία στα οποία θα διαφωνούμε και στα οποία θα διαφωνεί και το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο όμω κάνουμε σπάνια τελικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να προτιμάσουμε μία θέση διαπραγμάτευσης είναι σημαντικό να καταφέρουμε να προετοιμάσουμε τη θέση αυτή, τη διαπραγματευτική, βάσει τη οποία θα καταφέρουμε να συζητήσουμε στη συνέχεια και με το Συμβούλιο. Προσπαθούμε όμω και για πρώτη φορά να διερευνήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις νέε αρμοδιότητε που έχουμε πλέον ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίε απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Και προσπαθούμε μέσω αυτών να βελτιώσουμε την νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιλύσουμε κάποια υφιστάμενα πολιτικά και νομικά προβλήματα τα οποία εκκρεμούν για, πολλά, για πολύ καιρό. Έχουμε λοιπόν μια καταπληκτική ευκαιρία αύριο να καταφέρουμε να θεσπίσουμε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό και προοδευτικό πλαίσιο εξυγχρονισμού του εκλογικού συστήματος, εκλογικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και σαφώς ε, είμαι στη θέση σας να μιλήσω ακόμα και στις πολιτικές σας ομάδες και να παρουσιάσω περισσότερο τις ε, προτάσεις αυτές, καθώς θα βαδίζουμε προς την καταληκτική προθεσμία του Ιουνίου, της Ολομέλειας του Ιουνίου. Ευχαριστώ τον κύριο Νταφ. Έχω τρεις αγορητές. Ο κύριο Σέπφιλιν καταρχάς, ο κύριο Γκουαλτιέρη και ο κύριο Σταρκόσκη μετά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και στο παρελθόν θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφ. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία μαζί του Νομίζω ότι η Ολομέλεια του Ιουνίου ναι, όντως είναι και για μας μια ευκταία προθεσμία. Είναι καλό να παρατείνουμε την συζήτηση. Ο κύριος Σταφ βέβαια θα γνωρίζει όπως και εγώ ίδιος και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι ότι στην αρχή είχα την εντύπωση ότι υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί για τις διακρατικές αυτές λίστες, το διακρατικό συνδυασμό. Το να καταφέρουμε να έχουμε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο είναι πολύ καλό. Όσον αφορά τώρα τους ε, κλειστούς καταλόγους, την κλειστή λίστα, εγώ θέλω να είναι κλειστή λίστα όσο το περισσότερο για λόγους που σας είχα εξηγήσει στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες. Τον έχουμε ανοιχτούς καταλόγους, ουσιαστικά θα προμοδοτούσε περισσότερο τα μεγάλα κράτη γιατί θα επέτρεπε σε εκλογείς από τα μεγάλα κράτη να προωθήσουν περισσότερο τους δικούς τους υποψηφίους. Θεωρώ ότι κλειστοί κατάλογοι προωθούν περισσότερο τις μικρές ε, χώρες. Καταλαβαίνω βέβαια όλους αυτούς τους λόγους δημοκρατικής νομιμότητας φαίνεται πολλές φορές σε κάποιες περιπτώσεις ότι κάποιες λύσεις που προωθούνται σε δημοκρατικές μπορεί να μην φαίνονται τόσο ότι είναι δημοκρατικές. Ω προς τις μειονότητε, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και συμφωνώ απόλυτα ότι όντω θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τη σφαιρική εικόνα στη φάση αυτή και όταν φτάσουμε στη πραγματική φάση με το Συμβούλιο τότε θα πρέπει να μείνουμε περισσότερο στα επιμέρους σημεία. Όντως, το είπα στο παρελθόν, το ξαναλέω και τώρα, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος και οι διακρατικές αυτές λίστες θα μας επιτρέψουν πραγματικά να εκπροσωπηθούμε πολιτικά στο χώρο αυτό, να εκπροσωπήσουμε πολιτικά το χώρο αυτό. Έναν καθαρά ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος βέβαια θα χαίρει της άμεσης εκλογής από τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πολύ δυνατός σύνδεσμος ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και τους ψηφοφόρους. Το πώς θα λειτουργήσει όμως στην πράξη, με ποιο τρόπο, αυτό θα αποφασιστεί στο μέλλον. Όσον αφορά πάντω σφαιρική εικόνα και όσον αφορά την διαπραγματευτική μα θέση την οποία θα πρέπει εμεί να διαμορφώσουμε, πιστεύω ότι όντω τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μπορούμε εδώ να ακολουθήσουμε όντω να, τον κύριο Ντάφ και πιστεύω ότι όντω θα καταλήξουμε σε μια βελτίωση της νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ντάφ με τη σειρά μου γιατί ήταν και διατεθειμένος και να αντιπαρατεθεί αλλά και να συμβιβαστεί με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Δεν θα επανέλθω στα σημεία τα οποία επιλύσαμε στο παρελθόν. Θα επικεντρωθώ στα τελευταία σημεία που έθιξε. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχει διαγραφεί από τη συμβαστική πρόταση Α η μνήα τις ε, υποεθνικές ε, περιφέρειες, τις οποίες δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στη συνθήκη. Και εδώ θα ήθελα να δω μήπως θα έπρεπε να διαγράψουμε και αυτό που έχουμε στο άρθρο 3, δηλαδή να μην περιλαμβάνεται το στοιχείο που έχουμε στην τροπολογία υπαριθμών 4, διότι αφενός έχουμε την πράξη του 76 που αφορά το κατόφλι και δεν θα έπρεπε στο σημείο αυτό να αναφερόμαστε στις ε, περιφερειακές και τοπικές ε, αρχές στο σημείο αυτό. Για μας επίσης, καλώς έχει διαγραφεί η αναφορά στο σταυρό προτίμησης ε, στις εθνικές λίστες για τον ίδιο λόγο που τον έφερε και ο συνάδελφος Σέπφλιν και επίσης ευχαριστώ τον κύριο Νταφ διότι στο άρθρο 6 έχει διατηρήσει την ε, πολύ σημαντική αναφορά κατά την άποψή μου στις εκλογές χωρίς ε, δεσμεύσεις ε, θητείας για τους ευρωβουλευτές. Τώρα, για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες υπάρχει το ζήτημα που ήδη συζητήσαμε για το άρθρο 6α το οποίο προτείνω να αντικαταστήσουμε για τους καταδικασθέντες με οριστική απόφαση και θα πρέπει να δούμε λίγο τη διαδικασία του ποιος αποφασίζει και πώς αποφασίζει. Επειδή ακριβώς έχουμε μια νέα διαδικασία, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει να ισχύει με την έναρξη ισχύω. Επομένω, εδώ, ε, συγγνώμη, με την ημερομηνία των εκλογών. Επομένω, θα πρέπει ίσω να έχουμε αποφασίσει ήδη για την ημερομηνία των επόμενων ευρωεκλογών για τις ε, μειονότητες. Κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε να αναφέρονται οι εθνοτικές και οι γλωσσικές ε, μειονοτικές ομάδες να αναφερθούμε στο αρχικό κείμενο και να λέγεται απλώς ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών και των ε, μειονοτήτων. Ευχαριστώ στον κύριο Ντάφ που μας επιτρέπει να κάνουμε μια κατατμήματα ψηφοφορίας που κατά την άποψή μας είναι το πιο σωστό εδώ για την συμβιβαστική πρόταση J έχουμε ζητήσει να γίνει κατά τα ψηφοφορία για να μην αναφέρεται η αρχή της φθήνουσας ε, αναλογικότητας. Και αυτό προκύπτει από δύο στοιχεία. Πρώτον, πρόκειται για μία αρχή που ούτως ή άλλως από αυστηρά επιστημονική σκοπιά είναι δύσκολο να το καθορίσουμε. Επίσης δεν θα θέλαμε να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά που μας οδηγεί να θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι λίγο πολύ ένομο. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια πιο θετική αναφορά. Μία αναφορά ε, για ένα νέο μαθηματικό τύπο, τον οποίο θα πρέπει να ε, βρούμε. Και εδώ έχουμε και τις δικές μου τροπολογίες, ε, να δώσουμε δηλαδή ένα πιο θετικό τόνο στην έκθεση και να μην είμαστε τόσο επικριτικοί και αρνητικοί σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και λόγω των συζητήσεων που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την νομιμότητά του. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τις θέσεις μας, να ευχαριστήσω εκ νέου τον κύριο Ντάφ. Ευχαριστώ λοιπόν ο κύριο Σταρκόσκι. Well, Ευχαριστώ. Άντρου και συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που είχες. Θέλω να σου πω ότι το έχω σκεφτεί και το συζήτησα με πολλούς από ΜΚΟ και άλλες ε, οργανώσεις. Νομίζω οι πολίτες θα κρίνουν ε, το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο ως προς την αξία του, το, αν θα είναι ανοιχτό ή κλειστό. Υπάρχουν μερικά επιχειρήματα, δεν τα πιστεύω όλα, αλλά ε, εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Ε, ορισμένοι θεωρούν ότι ορίστε, δημιουργείτε καινούργιε θέσει για τους δικούς σας, για να βγουν οπωσδήποτε κάποιοι και να είναι σίγουροι ότι θα εκλεγούν. Και όταν είναι κλειστό το ψηφοδέλτιο είναι, έχει και κάποια ανοσία εντό εισαγωγικών ως προς την εθνικότητα, ε, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κρίνουν αυτό οι πολίτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε γνωστά ονόματα σε ψηφοδέλτια, όχι στα κόμματα και στους μηχανισμούς, αλλά στους πολίτες. Και αυτό δεν μας ενδιαφέρει η προβολή των πολιτικών κομμάτων. Δεν έχει κανένα νόημα να είναι ανοιχτή η κλειστή λίστα, αλλά αν χρειαστεί να το διαπραγματευτείς με το Συμβούλιο, να ξέρουμε ότι εκεί είναι το σημείο τριβής, από εκεί θα μας κρίνουν οι πολίτες. Και αυτό είναι το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο και αξία του. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση νομίζω. Ιδιαίτερα τη στιγμή που θα χρειαστεί να καθίσουμε και να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να τοποθετηθείς τώρα. Ξέρω ότι θα τα ξανασυζητήσει αυτά με το Συμβούλιο αργότερα. Ε, όχι το σύστημα DONT, να είναι πιο αναλογικό το link. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε, να μην είναι ταυτόχρονα παρόντες σε δύο ψηφοδέλτια. Τι θα γίνει όμως αν εκλεγεί κάποιος που συμμετέχει σε δύο ψηφοδέλτια, και στο εθνικό και στο υπερεθνικό. Θα θεωρηθεί ε, εκλεγής στη χώρα του, θα παραιτηθεί και θα περάσει ο πρώτος επιλαχών, θα θεωρηθεί εκλεγής με βάση το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Πώς το βλέπεις. Και στη συνέχεια, για το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο Είπε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πού ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Σε τέσσερα σημεία. Θα τα ψηφίσουμε ξεχωριστά ή όλο το συμβιβασμό. Δεν κατάλαβα. Σου μιλώ για τη συμβαστική τροπολογία L. Going, going to Ναι. Άρα θα ψηφίσουμε αύριο όλη τη συμβαστική τροπολογία. L. Ή 1, 2, 3, 4 ενημερωτικά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Το ΙΒ μάλλον είναι το ελληνικό κείμενο. Παρακαλώ. Ο κύριος Χέφνερ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Άντρου Ντάφ για την επιμονή του, την αιμονή του. Εδώ και καιρό παρακολουθεί αυτό το θέμα με μεγάλη μεθοδικότητα. Οι συζητήσει ε, τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες νομίζω βοήθησαν να οριμάσει το θέμα και να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα που μπορούν να δεχτούν ε, με μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα για τον τρόπο εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συμβαστικές τροπολογίες αυτό το τελευταίο που ρώτησε ο Ραφαέλ Τρασκόφσκι. Αν έχουμε δύο λίστες τώρα, δύο ψηφοδέλτια. Ένα που θα εκλέγει το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άλλο το συμπληρωματικό για την πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, την οποία επιθυμούμε. Αλλά εμείς πάντα ρωτούσαμε αν θα είναι επιπλέον. Ε, θα είναι 270, 251 ε, συν 25 ή αυτοί 25 οι βουλευτές, ευρωβουλευτές επικρατείας εντός εισαγωγικών θα είναι τμήμα των, 200, 751. Ναι, Ινίγκο, ξέρω ότι φρονείς εσύ να σας πω τι πιστεύω εγώ σε ορισμένα κρατημέλη ε, συζήτηση για διεύρυνση, αύξηση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολη. Και νομίζω ότι θα ήταν έξυπνη μια λύση που θα ε, λάμβανε υπόψη τα εξή δύο. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Αυτή η 25 να ε, είναι προς όφελος των μεγάλων κρατών γιατί έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγούν δικοί τους από ότι πολίτες μικρών κρατών. Επίσης και άλλους κινδύνους δεν το λένε πολύ συχνά, αλλά εγώ το βλέπω ότι ενδεχομένω θα ήταν και υπέρ των μεγάλων κομμάτων, όχι μόνο των μεγάλων κρατών. Αν λοιπόν κάποιος δεν θέλει η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στρεβλωθεί, ανοίγουμε ανοιχτό το μαθηματικό τύπο, αλλά κατά τα άλλα συμφωνούμε όλοι ότι η σημερινή κατανομή εδρών χρειάζεται επεξεργασία και αναθεώρηση και θα πρέπει να βρεθεί ένας μαθηματικός τύπος που να ακολουθεί ένα ενιαίο κανόνα και την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, αλλά να εφαρμόζεται με τρόπο ξεκάθαρο. Οπότε, εγώ τι λέω, να υπάρχει μια ρύθμιση που 25 που θα εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσμετρώνται στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, όχι επιπλέον ε, έδρες για τα κόμματα για τις χώρες, αλλά ο αριθμός εδρών αναχώρα που είναι γνωστός και περιορισμένος με βάση τη μαθηματική φόρμουλα ή το μαθηματικό τύπο. Λοιπόν, και ο αριθμός των εδρών που παίρνει ένα κόμμα να ε, προσανατολίζεται στο συνολικό αποτέλεσμα του και να έχουν επιλογή οι πολίτες να ψηφίζουν ένα βουλευτή, ευρωβουλευτή επικρατείας και ε, περισσότερους και μετά τους ε, εθνικούς, τα εθνικά τους ψηφοδέλτια. Αυτά. Ως πρόταση και δεν νομίζω ότι είναι τελείως άχρηστη αυτή η αντιπαράθεση. Τώρα, σύντομα για τα υπόλοιπα. Σε όλες τις τροπολογίες βλέπω εγώ βελτιώσεις σε ένα σημείο θεωρώ το θέμα ακόμα άλυτο. Αν έχουμε ενιαία φόρμουλα, ενιαίο μαθηματικό τύπο και στο μέλλον πραγματικά ε, να υπάρχουν σαφείς κανόνες, σε πόσους πολίτες αναλογεί μια έδρα, πόσες ψήφους θέλει κάποιος για να εκλεγεί, να είναι σαφής κανόνας, είπαμε για όλους ο ίδιο. Θα πρέπει να είναι η ίδια και η κλίδα καταμέτρησης στα κράτη-μέλη να είναι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου. Citizens λέει η συνθήκη και δεν λέει πουθενά κάτοικοι, residents. Είναι λάθος ο υπολογισμός. Καλά, ιστορικά μπορεί να εξηγείται και τεχνικά μπορεί να εξηγείται, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι αυτό ρυθμίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο αριθμός των πολιτών που δικαιούνται ψήφο είναι γνωστή, γνωστός και ο αριθμός των πολιτών. Και με μεταβατικές ρυθμίσεις μπορούμε να το κανονίσουμε προς το παρόν, ε, να μετρούν οι κάτοικοι, αλλά στο μέλλον οι ε, πολίτες πραγματικά, όχι μόνο εκείνοι που διαμένουν στη χώρα. Για να μην υπάρχει ε, αντίφαση στο ίδιο το νομικό κείμενο. Κατά τα άλλα χαίρομαι πάρα πολύ για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα συμφωνήσουμε, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Αυτά τα δύο σημεία είναι για μας αυτά που αξίζουν ακόμα συζήτηση και σκέψη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χέφνερ, ο κύριος Μπρόντς. Yes, uh, <clears throat> Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος ο οποίος θεωρεί ότι οι μαθηματικοί υπολογισμοί που γίνονται στις τρεις τελευταίες τροπολογίες είναι λίγο δύσκολοι. Φαντάζομαι ότι όταν χρειαστεί να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες αυτές στην Ολομέλεια δεν θα είμαι ο μόνος ο οποίος θα βρίσκει τη μαθηματική τους αν θέλετε κάπως δύσκολη. Στις τρεις αυτές λοιπόν τελευταίες τροπολογίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διατύπωση μόνο που θα περιλαμβάνει λέξεις και όχι μαθηματικά και κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να τις διαφοροποιήσουμε και ενδεχομένω και απλοί άνθρωποι σαν και εμένα καταφέρουν τότε να τις καταλάβουν και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα συμφωνήσουν μαζί μου και που δεν θα δυσκολευτούν όπως και εγώ στην Ολομέλεια. Ο κύριος Μενέντης ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Ντάφ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και καταρχάς ε, έχει κάνει αναζήτηση, έχει κάνει εξαιρετικό έλεγχο των εκλογικών συστημάτων και θα ήθελα να το συγχαρώ και για την προσπάθεια που έκανε να εξεύει τον κατάλληλο μαθηματικό τύπο. Δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε, χρησιμεύσε για κάτι. Χρησιμεύει στο εξή νομίζω. Ε, ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τούδε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνουμε την κατανομή των εδρών, μάλλον δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι έπρεπε να πάρουν περισσότερες ε, έδρες και κάποιοι άλλοι που έλεγαν ότι είναι ζημιωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν δίκιο όλοι αυτοί. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η συμφωνία που υπάρχει βάση της έκθεσης Λαμασούρου Σεβερίν είναι ένας ε, πολιτικός συμβασμός, μια πολιτική συμφωνία. Και νομίζω ότι εξαιτία αυτού θα είναι πολύ δύσκολο αυτή η πολιτική συμφωνία να υποκατασταθεί από άλλη και πολύ περισσότερο δύσκολο εάν αυτό το συνδέσουμε και με την ε, υπερεθνική λίστα, το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Το να προσθέσουμε τους 25 στους 751 ακούγεται πολύ δελαστικό, αλλά νομίζω ότι η εφαρμογή του στην πράξη θα είναι πάρα πολύ δύσκολη αν όχι και αδύνατη και θα υπάρξουν και ε, πολύ δύσκολες απόψεις να τις υποστηρίξουμε από πλευράς ε, της κοινή γνώμης. Ο κύριος Σέπφλιν είπε, τον οποίο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για τον τρόπο με τον οποίο κατήφθηνε το και σε όλο αυτό το θέμα, ε, ότι είμαστε υπέρ αυτού του υπερεθνικού ψηφοδελτίου. ε, ξανανοίγω αυτή τη συζήτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει σταυρός προτίμησης ε, σε αυτό το υπερηθνικό ψηφοδέλτιο. Εγώ είμαι υπέρ ε, του σταυρού προτίμησης, αλλά με έπεισαν και τα επιχειρήματα όλων αυτών που είπαν ότι ο σταυρός προτίμησης θα δημιουργούσε υποψίες ότι οι χώρες με, τις περισσότερες, ε, με τους περισσότερους ψηφοφόρους θα ήταν πιο ευνοημένες και θα μπορούσαν να επιλέξουν τους υποψηφίους τους στο ψηφοδέλτιο. αλλά υπάρχει και ο κύριος ε, Τρασκόσκη, ο οποίος είναι πολύ ικανός ε, και ε, μίλησε και με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και είπε ότι θα προτιμούσε να αποφύγει τις υποψίες αυτές που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για τις μεγαλύτερες χώρες, για να υπάρχει και αυτό το στοιχείο του να εκλέγονται οι καλύτεροι. Μου δημιουργήθηκαν λοιπόν αμφιβολίες για όλα αυτά που μόλις είπατε, διότι ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσω αυτού του υπερεθνικού ψηφοδελτίου να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή συνείδηση. Εάν όμως ε, προσπαθώντας να αναδυθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και να αποφύγουμε όλες αυτές τις υποψίες ότι το ψηφοδέλτιο αυτό θα είναι ε, αυτό που θα χρησιμοποιούν τα, οι μεγάλες πολιτικές ομάδες και οι μεγάλες χώρες και να δημιουργούμε νέες υποψίες από το πουθενά σημαίνει ότι έχουμε κάνει κακή διαπραγμάτευση ήταν κακό το προϊόν που αγοράσαμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι, να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερου πολίτε και να πιστεύουν οι πολίτε ότι πρόκειται για ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίου από μια πολιτική ομάδα με συγκεκριμένη ιδεολογική άποψη. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτείτε κι εσεί αυτό που είπατε και ίσω θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε από σήμερα μέχρι την ψηφοφορία στην Ολυμέλεια για να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφέ αυτό. Όπω σα είπα, κύριε Πρόεδρε, συμφωνεί απολύτω με τον κύριο Σέπφιλιν. Όσα είπα αντικατοπτρίζουν την άποψη τη ομάδα μα. Αύριο, όταν ψηφίσουμε, θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πείσουμε όλο το Κοινοβούλιο και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντάφο, ο οποίος είναι διατεθειμένος να μιλήσει με όλες τις πολιτικές ομάδες, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν επακριβώς την πρόταση και γι' αυτό ακριβώς δημιουργούνται και πάρα πολλές αμφιβολίες. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να το εξηγήσουμε σε όλους και καλό θα ήταν να συζητηθεί και να ψηφιστεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Επίσης κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι από τούδο και στο εξή, από αύριο δηλαδή που θα έχουμε κείμενο, επαφείται πλέον σε εμά ε, ως εκπροσώπων των πολιτικών μας ομάδων να εξηγήσουμε στους άλλους αλλά να τίνουμε και δίκο νους γιατί αυτοί, εμείς είμαστε αυτοί που θα ψηφίσουμε και θα πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε και τα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κύριε Νταφ ε, διότι κάνατε δουλειά επάξια αυτών που κάνουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Μαρτίνεθ πριν προχωράμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θέλουμε οι Ευρωπαίοι σε οποιαδήποτε πολιτική ομάδα και να ανήκουμε να έχουμε κοινού στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τέν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Άντριο, τον συνάδελφό μου, γιατί τόσο καλή δουλειά και για το ευρωπαϊκό του ιδεώδες σύντομα να πω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Χέφνερ για το πώς προσμερτώνονται αυτές οι έδρες των 25 βουλευτών επικρατεία. Στο Συμβούλιο θα είναι μεγάλα τα προβλήματα και από τη χώρα μου επίσης ε, αν προταθεί να αυξηθούν οι θέσεις ε, των Ευρωβουλευτών, ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν ταιριάζει με τους καιρούς όπου καλούμαστε να ε, είμαστε φιδωλοί. Και στη Γερμανία το μόνο που συζητάμε είναι ο μηχανισμό στήριξη και διάσωση του ευρώ. Το είπα και την περασμένη φορά. Ε, δυστυχώς είχαν φύγει συνάδελφοι. Έχουμε τεράστια προβλήματα εφαρμογής όλων αυτών και στα μάτια των πολιτών. Και η καλή ιδέα του υπερεθνικού ψηφοδελτίου και αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε για τους πολίτες μπορεί να διαστερβλωθεί και να μας γυρίσει μπούμεραγκ. Και σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να προτείνω το εξή. Πρώτον, δεν χρειάζεται ε, μεγάλη αλλαγή τη συνθήκη. Αν παραμείνουμε στις 751 έδρες θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα και το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν θα έχουμε τη συζήτηση με τις μικρότερες χώρες δηλαδή. Ότι δεν θα πρέπει να ε, παραδώσουν ε, καμία έδρα παραπάνω για να την πάρουν οι μεγάλες χώρες εάν αυτοί οι 25 ευρωβουλευτές επικρατείες συμπεριληφθούν του 751, ε, νομίζω θα ήταν καλύτερα. Ας πούμε, εάν με βάση ένα τέτοιο υπερεθνικό ψηφοδέλτιο εκλεγούν 7 Μαλτέζοι, που ε, θεωρώ απίθανο, θα μπορούσαμε να το εξισορροπήσουμε με μια άλλη κατανομή. Δηλαδή για τα πρώτα δυόμιση χρόνια της θητείας θα είχαμε ένα Μαλτέζο παραπάνω και στο υπόλοιπο ήμιση ε, θα άλλαζε θα παρέδιδε την έδρα του. Παρακαλώ να το σκεφτείτε και αυτό και να το έχετε υπόψη σας ως συμβαστική ε, λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Άντριο Νταφ, να μπω και εγώ σε αυτή την ιεροτελεστία. Ε, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η αιμονή του, η επιμονή του, η υπομονή του όλα αυτά τα χρόνια με μέθοδο να το φέρει μέχρι και την ψηφοφορία. Πραγματικά αξίζει να του το αναγνωρίσει κανείς αυτό. Τρεις παρατηρήσεις έχω. Το θέμα του υπολογισμού. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, αριθμό βουλευτών και τι γίνεται με τους 25 ε, ευρωβουλευτές επικρατείας, για να το πω έτσι. Αναγνωρίζουμε ευρωπαϊκή επικράτεια, εκλογική περιφέρεια Ευρώπη. Ε, τότε αυτοί δεν μπορούν να μπουν στα εθνικά ψηφοδέλτια. Εάν συνεννοηθούμε για μια υπερεθνική λίστα, ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, να το τηρήσουμε. Και καλούνται οι πολιτικές οικογένειες να λύσουν το θέμα αυτό στο εσωτερικό των κομμάτων με την κομματική τους δημοκρατία για να φτιάξουν αυτά τα ψηφοδέλτια πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό θα έλεγα στο όλο εγχείρημα και το πιο ενδιαφέρον και στο μέλλον γιατί είναι θέμα του μέλλοντος αυτό μπορεί να μην έχουμε καθόλου εθνικές λίστες, να έχουμε ε, μόνο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις ευρωεκλογέ να κατεβαίνουν στην αναμέτρηση. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά μακροπρόθεσμα και μάλιστα πολύ μακροπρόθεσμα θα ήταν ε, για μένα η μόνη δυνατή λύση. Να κατεβαίνουν στις ευρωεκλογέ μόνο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Και βέβαια θα πρέπει να κερδίσουμε και τους πολίτες αυτή την προσπάθεια των βουλευτών επικρατείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια μεταβατική περίοδο λοιπόν, μια προσωνή ρύθμιση και ένα συνδυασμό ευρωβουλευτών που θα εκλέγονται από εθνικά ψηφοδέλτια και από υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της ισότητας και δικαιοσύνης μεγάλων μικρών κρατών, μεγάλων μικρών κομμάτων. Στη δική μου πολιτική ομάδα η εικόνα είναι πολύ αντιφατική. Ε, και είναι επίμαχο το θέμα, δεν σας το κρύβω. Ε, και πώς θα εφαρμοστεί ε, η φθήνουσα αναλογικότητα, γιατί επικρατεί ένας κίνδυνος και ένας φόβος. Να μην εκπροσωπούνται τα μικρά κράτη, σωστά, ή τα μικρότερα κόμματα, τα μικρότερα ευρωπαϊκά κόμματα. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, και ένα τρίτο, συμφωνώ με την πρόταση να ε, παρατείνουμε την προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή τη στιγμή που θα ψηφίσουμε ε, στην Επιτροπή, να έχουμε ένα χρόνο να συζητήσουμε ε, το θέμα αυτό και στα κόμματά μας και στις πολιτικές ομάδες και στην κοινή γνώμη πριν πάμε στην Ολομέλεια. Δηλαδή από τη στιγμή της ψήφιση εδώ στην Επιτροπή μέχρι την ψήφιση στην Ολομέλεια να έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με επιχειρήματα στις πολιτικές ομάδες και στα κόμματα και στην κοινωνία. Και ένα τελευταίο. Ε, ακόμα μια σκέψη μόνο. Κάτι μου λείπει εδώ ακόμα όπως και στο παρελθόν για το δρόμο όπου θα ακολουθήσουμε και πού θέλουμε να πάμε. Εντάξει το κείμενο. Δεν περιγράφουμε που θέλουμε να πάμε, λέμε μόνο πώς θέλουμε να πάμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Eh, Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνείτε όλοι αύριο το πρωί να ψηφίσουμε, αλλά η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να γίνει τον Ιούνιο. Επειδή τα έχουμε επαναλάβει αρκετέ φορέ τα θέματα, πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντάφ γιατί μα πιέζει ο yes, um... Μάλιστα. για το ζήτημα της ε, ανοιχτή ή μη ανοιχτή ή κλειστή λίστας με προτιμησιακή ψήφο. Όντως το λέω ξεκάθαρα ότι ε, προτιμώ την ε, προτιμησιακή ψήφο ή μη ανοιχτή λίστας γιατί θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση και ουσιαστικά καταφέρνουμε να προσελκύσουμε περισσότερους ψηφοφόρους. Αν οι ψηφοφόροι έρθουν στις κάλπες και συνειδητοποιήσουν εκεί ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν κλειστή λίστα και ότι το μόνο το οποίο μπορούν αυτοί ως ψηφοφόροι να κάνουν είναι απλώς να βάλουν ένα σταυρό σε σύνολο υποψηφίων, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και δεν νομίζω ότι πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής στις ε, ευρωπαϊκές εκλογές. Και δεν νομίζω ότι ε, προωθεί πάρα πολύ την ενισχυμένη σχέση ανάμεσα στο ψηφοφόρο και το κοινοβούλιο. Ενώ αν μπορεί ο ψηφοφόρος να επιλέξει ανάμεσα σε κλειστό κατάλογο νομίζω ότι προφανώς θα προτιμήσει να, να, να, μπορεί να έχει αυτή την προτιμησιακή ψήφο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις και ότι θέλουν ουσιαστικά να προασπίσουν τα συμφέροντα μικρών μεγάλων κρατών. Να σας υπενθυμίσω ότι στόχος της υπερεθνικής λίστας ε, είναι να σπάσει αυτή η αυστηρή αν θέλετε σχέση ανάμεσα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη, τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει εδώ πέρα να μπορέσουμε να επιτρέψουμε μια πιο πλουραλιστική εκλογική διαδικασία. Εναπόκειται όμως ε, στην Επιτροπή και στα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν επ' αυτού. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προκαταβάλω οποιαδήποτε συζήτηση που θα γίνει για το σημαντικό αυτό ζήτημα, συζήτηση που θα γίνει μεταξύ μόν και του Συμβουλίου. Ο κύριος Γκουαλτιέρη και Άλλοι Ιταλοί συναδελφοί αναφέρθηκαν στο ζήτημα των πρώην καταδικασμένων οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό και στην Επιτροπή και αλλού και αν προβλέπετε τελικά κάτι τέτοιο, αν να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή αν δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν χαίρουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους όσοι δηλαδή έχουν καταδικαστεί για ένα σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, εφόσον λοιπόν επιβληθεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα αποτελέσει αρμοδιότητα εθνική, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συγκεκριμένα, να επιβάλλει τέτοια απαγόρευση στα, στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ε, Ένωσης. Αυτό θα αποτελούσε καταπάτηση της αρχής της επικουρικότητας και θα ερχόταν σε αντίθεση με την ε, πρακτική που ακολουθείται σε πολλά κράτη-μέλη. σε σχέση με την παρατήρηση του κυρίου Γκουαλτιέρη για την υφιστάμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι δεν συνάδει δηλαδή με την αρχή της φθήνουσας συναλλογικότητας ότι δεν συμμορφώνεται καταλήλως με την αρχή αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αντιταχθώ στην ομιμότητα του Κοινοβουλίου αυτού που εξελέγει ουσιαστικά πρωτού αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και πρωτού αρχίσει να ισχύει η νομοθεσία η οποία ορίζει την φθήνουσα αναλογικότητα. Καταλαβαίνετε ότι στη φάση αυτή προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την νομοθεσία αυτή. Υπάρχουν πάντως τουλάχιστον ε, πέντε περιπτώσεις όπου η σύνθεση του υφιστάμενου κοινοβουλίου τίθεται κατά της αυθήνουσας αναλογικότητας και το έχουν προσέξει αυτό και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σαφώς έχουν ε, ακουστεί επικρίσεις από το Γερμανικό μοσποδιακό Σταγματικό Δικαστήριο για το ζήτημα αυτό. Και όλες αυτές οι επικρίσεις ε, θα συνεχίσουν να υφίστανται αν εμείς δεν καταφέρουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό μέσω ενός μαθηματικού τύπου διαφανούς, δίκαιου, βιώσιμου. Αν συνεχίσουμε να γνωρούμε την ύπαρξη του προβλήματος, τότε το δικαστήριο αλλά και άλλοι φορείς τελικά θα έρχονται συνεχώς να μας επικρίνουν. Η απόψή μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ήπια αυτή αυτοκριτική όσον αφορά την υφιστάμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούστηκε επίση ένα ερώτημα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα DON και το σύστημα SANTLAG. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στο σύστημα SANTLAGU, τάσεται περισσότερο υπέρ των μειονοτικών κομμάτων. Είναι πιο αναλογικό και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται στη γερμανική εκλογική διαδικασία και σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τώρα τις διπλές υποψηφιότητες, η απάντηση προς αυτό είναι ότι ο εκλεγής ευρωβουλευτής αν τελικά έχει εκλεγεί τόσο στην διακρατική λίστα όσο και στην εθνική περιφερειακή λίστα, τότε θα πρέπει προφανώς να επιλέξει. Είτε δηλαδή να εκπροσωπηθεί μέσω της υπερεθνικής λίστας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να είναι ένας εθνικός βουλευτής. Εναπόκειται λοιπόν στο συγκεκριμένο άτομο να πάρει την απόφαση αυτή και προφανώς θα πρέπει να πάρει την απόφαση αυτή γρήγορα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να καλυφθεί η θέση η οποία θα μείνει κενή από την λίστα αυτή από την οποία θα αποχωρήσει. Το επόμενο λοιπόν άτομο που έπεται θα πάρει τη θέση του και αυτό το ζήτημα ενδεχομένω να μα απασχολεί στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Δεν έχει προκύψει πάρα πολύ πάντω στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή. Νομίζω όμω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέρο τη συζήτηση στο μέλλον. Τώρα, για το ζήτημα αν θα πρέπει να έχουμε 25 επιπλέον βουλευτές ή αν θα πρέπει αυτοί οι 25 επιπλέον να πάρουν τη θέση του στα πλαίσια των 751 η θέση της ε, Επιτροπής μας είναι να έχουμε 25 επιπλέον βουλευτές. Οι περισσότεροι έχουν ταχθεί πέρα αυτής της άποψης. Ο Ιγκο Μέντες Δεβίγκο έχει δίκιο. Το να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να συμφωνήσει με την ε, συμπερίληψη αυτών των 25 επιπλέον βουλευτών στην υφιστάμενη σύνθεση του Κοινοβουλίου θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να το πετύχουν ούτε καν με την ενθάρρυνση του Κοινοβουλίου. Γιατί και εμείς ουσιαστικά θα είμαστε διχασμένοι ανάμεσα στις ε, εθνικές αντιπροσωπίες και τα πολιτικά μας ε, κόμματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συνένεση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και τις εθνικές αντιπροσωπείες. Αν καταφέρουμε να πετύχουμε ένα υψηλό επίπεδο συνένεσης νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να εγκρίνουμε την θέση αυτή να έχουμε 25 επιπλέον βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προέρχονται από τη διακρατική εκλογική περιφέρεια. Ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητε μα μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχει αυξηθεί ο φόρτο εργασία, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και επιπλέον βουλευτέ θα βρισκόμαστε όλο και περισσότερο στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται για νέους βουλευτές οι οποίοι θα είναι δραστήριοι βουλευτές και οι οποίοι θα έρθουν να βοηθήσουν τους υφιστάμενους 750 με την δουλειά την οποία κάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι ε, πρέπει να πειραματιστούμε, αν μη τι άλλο, να πειραματιστούμε. Τη λέξη αυτή θα ήθελα να χρησιμοποιήσω με την ιδέα αυτή. Και απευθυνόμενος προς τους Γερμανούς, θα τους έλεγα ότι ε, το προηγούμενο κοινοβούλιο είχε 785 μέλη δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι εξωφρενικό να ζητάμε αυτή τη στιγμή 25 επιπλέον βουλευτέ και το λέω αυτό στου Γερμανού οι οποίοι πάντα ασχολούνται με τα οικονομικά. Ο κύριο ε, Μπόν αναφέρθηκε στην στο μαθηματικό τύπο. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί. Στην συμβαστική τροπολογία J, J, όντως προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για έναν και μόνο μαθηματικό τύπο, ότι χρειάζονται, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μαθηματικοί τύποι και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο. Εφόσον λοιπόν εγκριθεί και όπως πιστεύω ότι θα γίνει η συμβαστική τροπολογία Ι, τότε οι τρεις αυτοί προτινόμενοι μαθηματικοί τύποι θα καταπέσουν. Ο κύριος Σόλτς αναφέρθηκε στα μικρά κόμματα. Τα μικρά κόμματα αυτά χρειάζονται μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεποίθησης στα πλαίσια μιας διακρατικής εκλογικής λοιπόν περιφέρειας. Πιστεύω ότι θα τα πάνε καλά. Η Γκου, για παράδειγμα, θα μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να κερδίσει περισσότερη υποστήριξη σε χώρες όπου δεν έχει εκπροσώπους αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι έχετε Βρετανό από τη Βόρεια Ιρλανδία, ναι. Υπάρχει ένας βουλευτής. Πάντως, η λίστα της Γκουε θα μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει παντού σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, ε, καταλαβαίνετε ότι θα, μπορούς, θα μπορέσουν να αποφανθούν για τη δική σας την ε, λίστα ε, πάρα πολλοί άνθρωποι στον Ηνωμένο Βασίλειο, ότι βρίσκονται στην Αγγλία, είτε βρίσκονται στη Σκωτία, είτε στη Βόρεια Ιρλανδία. Εγώ προσωπικά δεν θα υποστηρίξω, αλλά θα υπάρχει μεγαλύτερη νόμιμη εκπροσώπηση υπάρχουν πάρα πολλέ πολιτικέ ομάδε, πολλά πολιτικά κόμματα τα οποία φοβούνται ότι θα πληγούν από το νέο αυτό σύστημα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν να θυγούν, ούτε θα τα πάνε αναγκαστικά άσχημα σε μια εκλογική διαδικασία, αν ισχύσει αυτή η υπερεθνική εκλογική περιφέρεια, η υπερεθνική εκλογική λίστα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε στην ιδέα αυτή μια ευκαιρία, να πειραματιστούμε με την ιδέα αυτή, να συζητήσουμε το Συμβούλιο και να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινώς ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. Εσ' αύριο είναι η ψηφοφορία, μετά από τις 10. Μετά τις 10 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ε, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ε, διοργανική συμφωνία για το κοινό μητρό διαφάνεια μεταξύ του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα συζητήσουμε από κοινού με το σημείο παριθμών 7 που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού μετά τη θέσπιση του κοινού μητρό διαφάνειας. Επειδή είμαι εισηγητή εγώ και θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί και το σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση πριν ακούσω τις παρατηρήσεις σας για το πώς έχει κατάσταση. Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της υποχρέωσης εγγραφής ε, στο Μητρό Διαφάνειας των ε, περιφερειών, επί παραδείγματι, των υποεθνικών ε, οργανισμών υποκρατικών. Έχουμε, έχουν κατατεθεί τροπολογίες και έχουμε καταλήξει σε ένα συμβιβασμό που ε, ελπίζω να διασκεδάσει όλες τις ανησυχίες και στη συμβιβαστική αυτή τροπολογία λέγεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εγγραφής στο Μητρό Διαφάνειας των ε, δημόσιων αρχών ε, περιφερειακού τύπου μόνο των υψηλών αντιπροσώπων. Δεν χρειάζεται να εγγραφούν ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, αλλά εάν υπάρχει αυτόνομος φορέας και δεν ε, ανήκει στις ε, αρχές ε, σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής. Αυτό θεωρούμε ότι διευκρινίζει όλα τα σημεία και το έχουμε συμπεριλάβει στο παράρτημα 1 που περιλαμβάνει τον κατάλογο όλων των οργανισμών και φορέων που μπορούν ή δεν μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στο, διαφάνιο, στο Μητρό Διαφάνειας. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόληση είναι το θέμα του υποχρεωτικού, της υποχρεωτικής εγγραφής στο Μητρό. Εγώ θα είμαι κατά σε τροπολογίες που θέλουν ως μελλοντικό στόχος ε, το Μητρό αυτό να είναι υποχρεωτικό. Το μητρό αυτό κατά την άποψή μου είναι ήδη υποχρεωτικό. Γιατί λοιπόν ε, παρερμηνεύουμε τον όρο υποχρεωτικός. Άλλο είναι η γενικευμένη υποχρέωση να εγγραφεί κάποιο, άλλο είναι το να πρέπει κάποιος να είναι εγγεγραμμένος εάν θέλει να συμμετέχει σε μια ομάδα πίεσης. Σε... Με άλλα λόγια, όποιος θέλει να επηρεάζει υπό την έννοια του ε, υποδεικνύει τα συμφέροντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρό Διαφάνειας. Υπ' αυτή την έννοια είναι υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρό Διαφάνειας αλλά δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε φορέας που δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις ε, με το Κοινοβούλιο και να έχει κάποια επιρροή ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρό Διαφάνεια. Κατά την άποψή μου λοιπόν ήδη είναι υποχρεωτικό το Μητρό διαφάνεια, όπως ακριβώς σας εξήγησα. Επομένως οι τροπολογίες και υπάρχει μια συγκεκριμένη τροπολογία που θέλει το μητρό διαφάνειας να λέγεται υποχρεωτικό μητρό διαφάνειας και μου δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, διότι θεωρεί ότι το μητρό διαφάνειας είναι υποχρεωτικό για οποιονδήποτε ε, θέλει να έχει ε, σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τροπολογίες οι οποίες λένε ότι ελπίζουμε ότι το μητρό θα γίνει υποχρεωτικό. Ήδη υποχρεωτικό είναι, κατά την άποψή μου και αυτή σας προτείνω και στο κείμενό μου. Επίσης υπάρχει και μία τροπολογία η οποία ουσιαστικά καλύπτει και κάποιες άλλες που ζητούν αλλαγή της συμφωνίας και άλλες που ζητούν τροποποίηση της συμφωνίας. Η συμφωνία έχει επιτευχθεί. Δεν ε, μπορώ να πω ότι θα είμαι αρνητικό σε τροπολογίες που ζητούν να γίνει κάποια δουλειά και να βελτιώσουμε λίγο τη συμφωνία. Και επίση υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίε κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι απαράδεκτε, διότι δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμφωνία. Ή θα τη δεχτούμε ή θα την απορρίψουμε, αλλά δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Αυτά από πλευρά μου νομίζω. Δύο είναι τα θέματα. Έχουμε καταρχά τη διοργανική συμφωνία και επίση την τροποποίηση που πρέπει να κάνουμε στον κανονισμό λόγω τη διοργανική συμφωνία. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει και το εξή. Αν πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία όπως υπάρχει, υπό την επιφύλαξη φυσικά και των ε, τροπολογιών που θέλουμε να κάνουμε εμείς ε, και τα όσα αναφέρονται στο αρχικό μου κείμενο, ή αν πρέπει να περιμένουμε, διότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας που έχει λάβει υπόψη και τα πρόσφατα γεγονότα που γνωρίζουν της ε, διαφθοράς ή της υποτιθέμενης διαφθοράς, μπορεί να κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε το θέμα, σα υπενθύμασα ότι πρόκειται για συμφωνία που αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά λοιπόν μια διοργανική εσωτερική συμφωνία, αφορά κάποιε πτυχέ, αλλά δεν μπορεί να αφορά την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου όσον αφορά τη διαφθορά, τη συμπεριφορά τρίτων προ το προσωπικό του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και άλλα τέτοια θέματα. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα και υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά δεν έχουμε καταλήξει στον τελικό στόχο της διαφάνειας. Πρόκειται για ένα βήμα προς τα μπρος, ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες, μία του συναδέλφου Νταφ και μία κάποιου άλλου μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, που πιστεύω ότι θα πρέπει να ενοποιηθούν για να εκφραστεί και αυτή η άποψη μου έχει δοθεί και ένα κείμενο με τρεις συμβιβαστική τροπολογίας. Τις έχω λοιπόν και γραπτός και σε μία συμβιβαστική τροπολογία έχει προσθεθεί ένα σημείο προκειμένου να έχουμε και τον απόλυτο συμβιβασμό εδώ. Έχετε λάβει κι εσείς το κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να ξαναδούμε τις τροπολογίες. Η πρώτη είναι η συμβασική τροπολογία Α που καλύπτει πολλές άλλες τροπολογίες και προσθέτει στο σημείο Β της έκθεσης για την έγκριση της συμφωνίας ότι δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή για εκπροσώπους που απαιτούν τμήμα της ε, διοίκησής τους λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό τους ρόλο ε, για τις ε, συνθήκες ε, στους παραγράφους 10, Β, 11, 12 και 13 και αυτό εδώ εκφράζεται και θα πρέπει να διευκρινιστεί λίγο καλύτερα στην επόμενη αναθεώρηση της συμφωνίας. Επίσης, εδώ προσθέτουμε και ότι ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δηλώσει και αυτή ότι συμφωνεί να γίνει περαιτέρω διευκρίνηση. Θα προσθέσουμε λοιπόν μια τελευταία φράση ότι η Επιτροπή δηλώνει και την ε, συμφωνία της, τη συμφωνή γνώμη της. Αυτό στη συμβαστική τροπολογία Α. Για τη συμβαστική τροπολογία Β τώρα, να σας το διαβάζω στα γαλλικά για το σημείο C του άρθρου 6, της παραγράφου 6, όπου αναφέρονται οι πιο σημαντικές πτυχές της συμφωνίας και, και λέει ότι το γεγονός ότι το Μητρό δημιουργεί διαφάνεια για τις ε, ποικίλε επαφές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ομαδοποιεί σε ξεχωριστά κεφάλαια εκπροσώπους ε, ιδιωτικών συμφερόντους, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους ε, δημοσίων αρχών και διακρίνει τον διαφορετικό ρόλο των ε, λόμπι και των επίσημων συνδιαλεγωμένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ λέει ότι ακόμα και η αυτόνομη εκπροσώπηση υπόκειται σε συγκεκριμένο νομικό καθεστώς. Επίσης έχουμε τη συμβαστική τροπολογία C που εισαγάγει μια νέα παράγραφο και λέει το εξής. 6α το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι εφαρμοστέοι κανόνες για τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών και των οργανώσεων που ε, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους εξυπηρετούν τα δημόσια συμφέροντα και σχετίζονται ε, στους συνταγματικούς ε, κανόνες τους ε, και στα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να είναι πανομοιότυπες με αυτές που εφαρμόζονται για τους εκπροσώπους συγκεκριμένων συμφερόντων και θεωρεί επίσης ότι η πρόσκληση να εγγραφεί κάποιος αφορά οργανισμούς ε, δημοσίου συμφέροντος και δεν θα πρέπει να αφορά οργανισμούς που έχουν αυτόνομα καθεστώς, ε, και, αλλά όχι και τις ε, δημόσιες αρχές. Ο κύριος Γκρέτ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα ενδιάμεσο στάδιο δεν έχει κλείσει το θέμα της διαφάνειας και δεν θα πρέπει να ε, συγχαίουμε αυτή την προσπάθεια με την ομάδα εργασίας ε, του Προεδρείου. Μας είπε πρόσφατα και η κυρία Γόλης ότι αποφασίστηκε στο Στρασβούργο να τον αναλάβει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αυτό και ο κύριος Κασίνη με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε ένα κείμενο και ε, είναι τώρα αυτό το κείμενο και μπορούμε να το υπερψηφίσουμε ή να το καταψηφίσουμε. Εγώ είμαι υπέρ της υπερψήφισης, έχουν γίνει συμβασμοί και πάλι είναι, δεν είναι ο τελικός προορισμός, είναι μια ενδιάμεση φάση. Οι τροπολογίες 37 και 38 είναι απαράδεκτες. Ε, στην έκθεση και χαίρομαι που βρήκαμε ένα συμβιβασμό και για τις ε, αντιπροσωπείες των ε, ΟΤΑ. Υπάρχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν περιφέρειες με συνταγματικό χαρακτήρα και δυνατότητα και αρμοδιότητες και εξουσίες κρατικού τύπου. Ελπίζω σύντομα να ε, έχουμε πλέον υποχρεωτικό μητρό και επίσης ένα κοινό μητρό με το Συμβούλιο. Και τα τρία θεσμικά όργανα να μπουν. Μπορούμε να το έχουμε αυτό. Δεν είναι αντικείμενο της παρούσης έκθεσης, αλλά είναι ο τελικός στόχος και όχι ε, Κάθε ομάδα επισκεπτών, κάθε ομάδα επισκεπτών που έρχεται εδώ αναφέρει αυτό το θέμα της διαφάνειας. Και δυστυχώς Είχαμε και αυτά τα περιστατικά στο Κοινοβούλιο που ήταν βέβαια μηχανογραφίες και παγίδες, αλλά ε, ισχύει για όλους και το βρίσκουμε όλοι μπροστά μας. Μας ρωτάνε και δυσάρεστα και τους λέω ότι 99% των συναδέλφων είναι αξιοπρεπείς και έντιμοι άνθρωποι. Αλλά θα πρέπει να μπει και αυτό το μητρό ε, μπροστά. Είναι ενδιάμεσο ο προορισμός, δεν είναι ο τελικός προορισμός αυτός. Ε, θα το υπερψηφίσουμε επιτέλους για να πάρει μπρος αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέφνερ. Εγώ μίλησα μόνο για τα ουσιαστικά σημεία, αλλά υπάρχουν και άλλε τροπολογίε για τι οποίε έχω εκφράσει την άποψή μου και τι οποίε θεωρώ δευτεροβούση σημασία. Δεν έχουν σχέση με τα θέματα τα οποία ανέφερα, γι' αυτό και δεν τι ανέφερα. Ο κύριο Χέφνερ. Ναι, και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο ε, για τα σημαντικότερα, ουσιαστικότερα θέματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ε, και αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Κασίνη, για την έκθεση αυτή και για τις συμβαστικέ τροπολογίες που προτείνετε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρότε. Αυτό είναι ένα βήμα ακόμα προς το τελικό μας προορισμό για μεγαλύτερη διαφάνεια και το βήμα αυτό χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μας ακολουθεί το Συμβούλιο, μόνο η Κομισιόν θα ήταν πολύ καλύτερο και για το ίδιο το Συμβούλιο και για μας να κάναμε και τα τρία θεσμικά όργανα το βήμα αυτό από κοινού. Για το θέμα τώρα του δεσμευτικού ή όχι χαρακτήρα. Συμφωνώ ε, στο εσωτερικό της λογικής που επελέγει και της νομικής βάσης τώρα. Είναι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση. Αν θέλουμε όμως υποχρεωτικό μητρό θα μπορούσαμε να βασιστούμε στο άρθρο 352 που επισύρει και κυρώσεις, διότι για μας το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα κυρώσεων. Αν είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό, όποιο το παραβαίνει δεν παθαίνει τίποτα. Απλώ δεν του δίνουν badge, δεν του δίνουν κάρτα εισόδου στο κοινοβούλιο. Αλλά αυτά που ενδιαφέρουν του πολίτε οι συζητήσει δεν γίνονται πάντα στο κοινοβούλιο, γίνονται και εκτό. Και πολλοί μπορεί να μπαίνουν ε, με άλλη κάρτα εισόδου δεν είναι ανάγκη να έχουν το badge του λόμπι, μπορεί να έχουν κάρτα επισκέπτη, ημερήσια. Εμείς λοιπόν καταχωρούμε ε, σε ένα μητρό ποιος μπαίνει στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένα τα λόμπι να δηλώνουν τις δραστηριότητές τους και τις επαφές τους με τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, η τέχνη του εφικτού. Ε, είπαμε, στα πλαίσια του εφικτού είναι πολύ καλή η συμφωνία και η τροπολογίες ε, συμβαστικές. Έχω κάνει σε δύο σημεία τροπολογίες, το ανέφερα το ένα είναι αυτό το ε, δεσμευτικό και το υποχρεωτικό και το άλλο αναφέρθηκε επίσης που είναι τις αντιπροσωπείες τοπικών κυβερνήσεων που είναι οντότητες με νομοθετικές εξουσίες Υποκρατικέ. Δεν μπορούν να θεωρούνται σίγουρα ως ομάδες πίεσης ή ο πρώτος τυχόν λομπίστα. Χαίρομαι που δεχτήκατε αυτές τις τροπολογίες και το καλωσορίζω. Και μπορούμε εμείς να πούμε ότι σε ό,τι μας αφορά έχει καλυφθεί το πρόβλημα. Αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό συζήτησα με την Επιτροπή και η πρώτη αντίδραση ήταν ε, έκπληξη και δεν καταλάβαιναν τι ζητούσα, γιατί μου λένε εδώ μέχρι και εκκλησίες πρέπει να δηλώνονται. Τι θες εσύ με τα κρατήδια. Ε, εγώ πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Μπορεί κάποιος να είναι ε, μέλος σε μια εκκλησία ή να μην είναι πιστός ή να βγει από την εκκλησία. Και είναι και πολλές οι εκκλησίες. Δεν το βάζω στο ίδιο επίπεδο, αλλά μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο Volvo, BMW ή στη Microsoft ή open source τα προγράμματά μου. Όλα αυτά είναι πράγματα που μπορώ να τα αποφασίζω κατά συνείδηση και το θεωρώ θεμητό ομάδες πίεσης που εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα να καταγράφονται. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω αν είμαι μέλος της Βαβαρίας ή της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Όταν είμαι πολίτης ε, έχω αυτό το καθεστώς, η μοίρα μου είναι να είμαι σε αυτό το κρατήδιο και δεν ισχύει μόνο στη Γερμανία αυτό, αλλά κυρίως στη Γερμανία που είναι αμοσπονδιακή χώρα. Ε, μεγάλο τμήμα της ε, κρατικής κυριαρχίας εκχωρείται προς τα κάτω ε, στα αμόσπονδα κρατήδια και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Αυτοί που εκπροσωπούν εδώ τα κρατήδια αυτά είναι τμήμα της διοίκησης, είναι υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε στα λόμπι. Το θεωρώ τελείως ανάρμοστο και ε, έχω πραγματικά παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που δεσμεύτηκαν απέναντί μου προσωπικά, ότι το κατάλαβαν και θέλουν να το αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το δηλώσει και δημόσια. Εδώ να γραφεί στα πρακτικά ή σε μια επιστολή. Γιατί δεν αρκεί να στο λέει κάποιο υπάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το καταλάβαμε ότι είναι διαφορετικό αυτό και το Κοινοβούλιο το γράφει στην έκθεσή του με την πρόταση του Πρόεδρου κ. Καζίνη, αλλά το δηλώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το κατάλαβε και ότι ισχύει και μέχρι την επόμενη αναθεώρηση και αναδιατύπωση της συμφωνίας θα το διατηρήσουμε έτσι. Παράκληση θερμή και πήγουσα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαμπρινίδης. Thank you, Chairman. Um, uh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την Προεδρία του κύριου Μπούζεκ θα γίνει αύριο. Η Νταϊάννα Γόλης και ο υποφαινόμενος θα συμμετέχουμε στην ομάδα αυτή ως αντιπρόεδροι. Και υπάρχουν ε, δύο σημαντικά σημεία. Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας των Ευρωβουλευτών και προτάσεις προς αυτό και αναθεώρηση του, κώδου, του κώδικα συμπεριφοράς των ε, εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω μία-δύο ερωτήσεις. Η διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει ξεκάθαρα έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους ε, ομάδων συμφερόντων. Λέγεται ξεκάθαρα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Παράρτημα 10 συγκεκριμένα, το οποίο έχει αντικατασταθεί από το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας. Το ερώτημά μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι η ομάδα εργασίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να αναθεωρήσει τους κανόνες αυτούς Κατά την άποψή σας, πιστεύετε ότι έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει το κείμενο μόνο για, το σκο... για σκοπούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά δηλαδή τη διοργανική συμφωνία, γιατί αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε τουλάχιστον σε σχέση με τη συμπεριφορά των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων, φαίνεται ότι εμείς σιωπούμε. Φαίνεται ότι έχουμε μια ομάδα εργασίας η οποία δεν τοποθετείται επ' αυτού. Δεύτερο τώρα ερώτημα. πώς αντιμετωπίζεται όντω τα ομόσπονδα κρατήδια. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τι θα γίνει όμως με τους ε, εκπροσώπους εκείνους που ε, δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από τρίτη χώρα. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την διπλωματική αυτή εκπροσώπηση, δηλαδή διοικητική υπάλληλη από τρίτες χώρες. Η Διοργανική Συμφωνία προβλέπει κάτι γι' αυτό ξέρω ότι η τροποποίηση της ε, νομοθεσίας είτε μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας την οποία εγκρίνουμε είτε ε, μέσω άλλων νομοθεσιών εκπροσωπούνται τέλο πάντων τα συμφέροντα των τρίτων αυτών χωρών μέσω των διπλωματικών αντιπροσωπιών τους, μέσω των πρεσβειών κτλ. Δεν πρόκειται όμως για λομπίστες, για εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, δεν υπάρχει αυτή η χρηματική εμπορική διάσταση, αλλά προσπαθούν να πειράσουν ουσιαστικά τη στάση των Ευρωβουλευτών και να τροποποιήσουν τρόπον την κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να καταχωρούνται λοιπόν ή όχι στα πλαίσια της οργανικής αυτής συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Τέιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για τις συμβαστικές τροπολογίες, ιδιαίτερα για τους εκπροσώπους ε, των ε, Μόσπονδων κρατηδίων γενικά των δημοσίων διοικήσεων. Είναι λοιπόν αυτή μια συμφωνία πλέον ε, που επετεύχθη, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να μας το δηλώσει τώρα, γιατί το λέει και η τροπολογία, ότι στην επόμενη διατύπωση θα διευκρινιστεί η συμφωνία. Δεν μπορείτε να το διευκρινίσετε από τώρα. Να βγάλετε τις εκπροσωπήσεις ε, των κρατηδίων. Άκουσα ο κύριος Χέφνα να λέει ότι να βάγισαν οι συνομιλίες. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να το δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε αναθεώρηση τη συμφωνία, να σβήσουμε δύο λέξει. Πέντε λεπτά και τελείωσε η υπόθεση. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να περιμένουμε. Και η Διαπραγματευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνεί. Και το μπαλάκι τώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παράρτημα 1 δεν μπορείτε να σβήσετε αυτέ τι δύο λέξει. Αυτά. Ερώτηση προ την Επιτροπή. Να μα εξηγήσει τι συμβαίνει. Να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Χέφνερ, ο οποίος θέλει να απαντήσει στην προηγούμενη. Ε, δεν θέλω να παραμείνει παρεξήγηση στο χώρο. Εγώ έκανα συνομιλίες και είπα στην αρχή προσέκρουσα σε έλλειψη κατανόηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν είχαν αναγνωρίσει το πρόβλημα. Στο τέλος όμως δεσμεύτηκαν ρητά να αλλάξουν αυτή τη διατύπωση με τον τρόπο που πρότεινε και συμβαστική τροπολογία ο κύριος Κασίνη. Αυτό μου το διαβεβαίωσαν προσωπικά και προφορικά. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να τους το προσάπτω. Ήταν εμπιστευτική η συζήτηση και σας το αναφέρω, αλλά θέλω επίσημα να το δηλώσει δημόσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γραφεί και στα πρακτικά. Ευχαριστώ, κύριος Ευχαριστώ. Ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Λαμπρενίδη. Γιατί και στην εργασία που πρέπει να επιτελέσει τα πλαίσια της νέας αυτής ομάδας εργασίας. Γενικότερα η Επιτροπή θεωρεί ότι η διοργανική συμφωνία είναι καλή με την παρούσα της μορφή, αλλά σε ορισμένες ε, περιπτώσεις δεν είναι αρκετά στεναρή. δεδομένης της αύξησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεδομένου του όλου κλίματος που υφίσταται, όπου ζητάμε ένα πιο ανοιχτό σύστημα διακυβέρνησης και ότι Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τον εγχείρημα αυτό τώρα. Ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα το διαπραγματευόμαστε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τον εγχείρημα αυτό και φαίνεται ότι υπάρχουν πλέον πολλοί οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την τροπολογία 30, στην οποία αναφέρομαι στην ε, οδηγία του legislative footprint, του νομοθετικού αποτύπωματος και που προσπαθώ να δω αν το Προεδρείο θα μπορούσε να επινοήσει ένα σύστημα βάσει του οποίου οι ευρωβουλευτές και ιδίω οι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να καταγράφουν τις επαφές τις οποίες έχουν με καταχωρημένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Ξέρω το ζήτημα αυτό είναι ευαίσθητο και ξέρω ότι θα είναι πολύπλοκο να συμφωνήσουμε επ' αυτού για μια διαδικασία τέτοια. Νομίζω όμως ότι αξίζει να το προσπαθήσουμε. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα υποστηρίξει την τροπολογία μου αυτή. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει να μιλήσει και ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν θέλει το λόγο μπορεί να παρέμβει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά τώρα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής θα μπορούσα να ε, Προτείνω τρία πράγματα υπόψη σας. Το πρώτο. Διαπιστώνω ότι μιλάτε για λόμπι για όλους εκείνους που θα πρέπει να καταχωρούνται. Βεβαίως, εμείς αποφύγαμε σε όλο το κείμενο να βάλουμε τη λέξη λόμπιστ. Γιατί, εάν το κείμενο συμπεριλάβει βέβαια και σε κάποιο βαθμό ε, ρυθμίζει τις σχέσεις που ε, έχουμε με τα λόμπι. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά αφορά και άτομα και οργανώσεις που συμμετέχουν στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Ακριβώς για να απαντήσουμε στην ανησυχία κάποιων οργανισμών που είναι εταίροι μας στις διάφορες διαδικασίες και δεχόμαστε ε, τη διαφάνεια εάν δεν θεωρούνται όμως λόμπι. Γιατί δεν υπάρχει και ορισμός αυτού. Οπότε για να γραφτεί, το να γραφτεί κάποιο δεν σημαίνει ότι έχει την ετικέτα λόμπι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι το μητρό αυτό που καταγράφει μόνο λόμπι. Στη συνέχεια είναι δύο τα άρθρα που θα πρέπει να τα βλέπουμε από κοινού και να τα εφαρμόζουμε από κοινού. Το πρώτο είναι το άρθρο 9, το οποίο έχει και μία υποσημείωση που λέγει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, διεθνών οργανισμών και οι πρεσβείες και οι διπλωματικές αποστολές δεν αναμένεται ή δεν απαιτείται να καταγράφονται. Σε μια ομοσπονδιακή χώρα όπου ε, έχουν εκχωρηθεί προς τα κάτω σε οντότητες υποκρατικές εξουσίες, στη δική μας ερμηνεία χωράνε εδώ. Δεν ισχύει μόνο για τα Λέντερ, για το ομόσπονδα κρατήρια στη Γερμανία. Αυτό μπορεί να ισχύει για την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που ε, έχουν τέτοιες περιφέρειες και άλλες χώρες. Το άρθρο 10 υπό παράγραφος Β ορίζει την αρχή ότι ότι οτιδήποτε ισχύει ε, εκεί ε, κατά αναλογία η μουτά της μουτάντης επεκτείνεται. Όταν έχει κάποιος μια δραστηριότητα που απορρέει από τη συνθήκη δεν εμπίπτει στον τομέα του Μητρώου. Δηλαδή, οποιασδήποτε δραστηριότητες των δημοσίων αρχών, ε, ανεξαρτήτως επίπεδου, που ε, αναλογούν σε δραστηριότητα που απορρέει από τη συνθήκη, είναι εκτός πεδίου εφαρμογή του Μητρώου. Γι' αυτό, κατά την άποψή μας, το κείμενο καλύπτει ε, αυτή την περίπτωση και προστατεύει αυτό που σας ενδιαφέρει. με αυτή την ε, ερμηνεία που μόλις σας είπα. Ο κύριος Χέφνερ εκτός μικροφών. I Κατανοώ την ερμηνεία σας, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί και πρέπει να διευκρινιστεί. Γιατί λέτε ότι κράτη-μέλη σημαίνει επίσης περιφερειακές αρχές και ούτω καθεξής. Και γιατί να μην το πούμε λοιπόν αυτό, διότι έχει δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις και γνωρίζω ότι κάποια από τα προβλήματα προέκυψαν περισσότερο από την έκθεση και όχι από το αρχικό κείμενο, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και θα πρέπει να υπάρχει και συνέπεια μεταξύ της έκθεσης και της συμφωνίας ε, αυτής καθεαυτής. Πρόεδρε, συγγνώμη, θέλω να πω κι εγώ. Καλύτερα να ζητάτε το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ναι ήθελα να πω το εξής. το έξι λατινικό, υποπαράγραφος, σε γραφεία εκπροσώπησης, ίσως θα βάλετε και εκεί υποσημείωση στο τέλος, τα γραφεία εκπροσώπησης δεν είναι γραφεία εκπροσώπησης ομόσποδων κρατηδίων, περιφερειών κτλ. Δεν είναι οι αντιπροσωπείες. Μιλάτε για γραφεία αντιπροσωπιών γιατί η αντιπροσωπεία ενός κρατηδίου θεώρησε ότι την αφορά. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Βάλτε και εκεί καμιά υποσημείωση. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κάνω μια απόπειρα να ολοκληρώσω, διότι έχουμε και συνεδρίαση συντονιστών αργότερα. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριο Λαμπρινίδη για άλλη μια φορά και μετά ο κύριο Γκρέτε. Και μετά θα ολοκληρώσω τι παρεμβάσει. Uh, no, Ξαναπέρνω το λόγο σε σχέση με αυτά που είπε ο Άντριου Νταφ που απαντούν εν μέρη το ερώτημά μου. Αν πάρουμε την τροπολογία του Άντριου, τότε όντως η τροπολογία αυτή έχει σχέση με την εντολή της ομάδας εργασίας, δηλαδή ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να είναι πιο διαφανείς οι ευρωβουλευτές και ενδεχομένως να έχουν και αυτό το περίφημο αποτύπωμα το νομοθετικό. Πρέπει όμως η ομάδα εργασία πρώτα να συνεδριάσει και μέσω συστάσεων να συνταχθεί και η έκθεση στην Επιτροπή αυτή. Αν γίνουν τα πράγματα αντίστροφα, τότε μπερδευόμαστε και ουσιαστικά θα έχουμε μια έκθεση τη Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων, Συνταγματικών με θεμάτων για το ζήτημα αυτό και στη συνέχεια η ομάδα εργασία θα πρέπει να κάνει ακριβώ την ίδια εργασία. Εσεί πρέπει να αποφασίσετε αυτή τη στιγμή πώ θα κινηθούν τα πράγματα. Ενδεχομένω να είμαστε λίγο αργά πια στο χρονικό περιθώριο το οποίο προβλέπετε. Δεν ξέρω πάντω αν οι δύο αυτέ οι δύο αυτοί φορεί αντιτάσσονται ένα στον άλλον. Είδα την υποσημείωση, χαίρομαι πολύ για αυτήν. Πιστεύω ότι δεν, μπορούν, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τις υποσημειώσεις περισσότερο. Απευθυνόμενος πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι αν είσαι στον κατάλογο αυτό και δεν είστε αναγκαστικά από μία ομάδα συμφερόντων, όταν είστε όμως στον κατάλογο αυτό σημαίνει ότι προσπαθείτε να επηρεάσετε με τον έναν τον άλλο τρόπο την κοινοτική νομοθεσία. Επομένως, αν προσθέσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες ε, εκ των πραγμάτων επηρεάζουν την ε, κοινοτική, τότε θα είναι λογικό να μην μπουν στον κατάλογο. Οι ξένες όμως κυβερνήσεις που δεν έχουν ε, ως βασικό στόχο να, έχουν, να παράγουν κοινοτική νομοθεσία, όταν εμπλέκονται και πειράζουν τελικά τη δική μας νομοθεσία, τότε θα πρέπει και αυτές να μπουν στο μητρό το να μπουν στο Μητρό δεν τις εξομοιώνει με λόμπι, θα είναι απλώς εξωτερικοί παράγοντες που προσπαθούν να, βοηθ... επηρεάσουν την κοινωτική νομοθεσία. Ενδεχομένως οι παρατηρήσεις μου αυτές πλέον έρχονται πολύ αργά, μπορούν να εξεταστούν πάντως στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι, θα έλεγα να το κάνουμε εξή απλούστατα, να μπει και το Συμβούλιο μέσα στο Μητρό και να έχει και επιρροή, να είναι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να μπορεί να τα διαπραγματεύεται. Να έρθει και το Συμβούλιο λοιπόν και να διαλύονται τέτοιες παρεξηγήσεις, γιατί είναι μέλη του Συμβουλίου αυτή. Ωραία, να κάνω μια απόπειρα να απαντήσω εντάχει στι ερωτήσει και στι παρατηρήσει σα. Καταρχάς, να πούμε ότι το θέμα του κώδικα δεοντολογίας, ε, γιατί κάποιος το είπε αλλά το ε, υπενθυμίζω, υπήρχε κώδικας δεοντολογίας, υπάρχει τώρα το παράρτημα 10 που είναι ένας νέος ε, κώδικας δεοντολογίας και περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Υπάρχουν κυρώσει, σαφώ υπάρχουν κυρώσει και είναι διαβαθμισμένε. Υπάρχουν 10 τύποι κυρώσεων και είναι ανάλογε τη παράβαση που γίνεται ε, χρειάζεται η νέα συμφωνία για να το εμπλουτίσουμε ή να το τροποποιήσουμε. Υπάρχει όμως. Για τη διπλωματική εκπροσώπηση τα ακούσαμε, δεν θα προσθέσω εγώ τίποτα. Εξαιρούνται οι διπλωματικές ε, αντιπροσωπείες από το Μητρό. Και εγώ συμφωνώ με τις δύο τροπολογίες και μάλιστα θα ήθελα να προτείνω να τη συμφωνήσουμε από κοινού με τον κύριο Ντάφ και τον άλλο συνάδελφο που παρουσίασε την τροπολογία υπαριθμό 3 νομίζω, διότι πρόκειται για ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Εμείς το επεκρίνουμε αρκετά γιατί δεν αρκεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε. Και υπάρχει μια τροπολογία που Ντάφ και που ζητούν από το Προεδρείο να σκεφτεί ένα σύστημα βάσει του οποίου ακόμα και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να εγγράφουν στο Μητρό τα ονόματα ανθρώπων που κάνουν ε, προτάσεις και να υποδοκνύονται αυτοί στην τελική έκθεση σε μια υποσημείωση λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων ήρθαν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση του συγκεκριμένου κειμένου. Εγώ προσωπικώ συμφωνώ αρκετά παρά το γεγονός ότι είναι πολύ περίπλοκο. Δεν είναι τόσο απλό, πολύ εύκολα το λέμε, πολύ δύσκολα το υλοποιούμε. Τώρα, τι θα πρέπει να σημειώνουμε, να σημειώνουμε μόνο αυτά τα οποία γίνονται μέσω ε, ομάδων συμφερόντων που είναι γεγραμμένοι στα Μητρώα ή και αυτοί οι οποίοι συναντούν τους ευρωβουλευτές αλλού εκτός Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποδεικνύουμε στην τελική έκθεση κάτι το οποίο υποστηρίζω μόνο τα ονόματα αυτών που προσέγγισαν τον εισηγητή ή και τους κοιόδης εισηγητές ή όλους τους ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου και πώς θα τα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με την ιδέα, θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και εμεί ω Επιτροπή, θα προσπαθήσει να το κάνει και η ομάδα εργασία, η οποία ομάδα εργασία, κατά την άποψή μου, έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα. Εγώ ειλικρινώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει εδώ διάσταση απόψεων. Εμεί ετοιμάζαμε ένα μητρό διαφάνεια, αρκεί προ το παρόν, υπάρχουν κυρώσει και υποχρεώσει και για τους ευρωβουλευτές και για τους ε, λομπίστες και τους εκπροσώπους συμφερόντος. Η συμφωνία δεν αναφέρεται σε λομπίστες, αναφέρεται σε οργανώσεις και πρόσωπα που θέλουν να συνεισφέρουν. Διότι δεν είναι πάντα κακή συνεισφορά. Η επιρροή στα Ιταλικά έχει κακή ε, ε, έννοια, έχει και μια κακή απόχρωση. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις ε, και να υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς τη διαφάνεια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήδη έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Σαφώς πρέπει να γίνουν και τα επόμενα και η ομάδα εργασίας κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει κατά νου ότι τα όσα συνέβησαν που είναι πολύ αρνητικά δεν οφείλονται σε άτομα τα οποία ήταν πραγματικά εκπρόσωποι συμφερόντων. Ήταν δημοσιογράφοι που παρίσταναν τους ε, εκπροσώπους συμφερόντων. Επομένως υπάρχει και η ευθύνη αυτού που πράττει. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα του ευρωβουλευτή. Υπάρχει και ένας τρίτος ο οποίος έρχεται σε επαφή με έναν ευρωβουλευτή και προσπαθεί να το διαφθείρει. Και αυτό δεν το κάνει μόνο στο κοινοβούλιο. Μπορεί να το κάνει και στο σπίτι του και στο δρόμο, σε ε, ε, ένα λεωφορείο. Υπάρχει λοιπόν λόγος να υπάρχει ένα μητρό διαφάνειας Και θα πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να έρθουμε σε επαφή με τα ε, θεσμικά όργανα για να κάνουμε τις επαφή μας. Και εδώ υπάρχει και διαφορά μεταξύ ε, εκπροσώπησης οικονομικών συμφερόντων αλλά και ιδεών που μπορεί να μην έχουν ε, απαραίτητα οικονομικό χαρακτήρα. Με αυτά λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία αύριο. Νομίζω ότι υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη σύγκληση απόψεων που θα φανεί και στην ψηφοφορία από εκεί και πέρα ε, θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν. Για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες θεωρώ ότι υπάρχει συμφωνία. Ο καθένας τώρα στις υπόλοιπε τροπολογίες θα εκφράσει την άποψή του αναλόγως. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο η γνωμοδότηση Μέσερ Σμιτ για την ε, Επιτροπή Νομιθετικών ε, ε, Νομικών Υποθέσεων έχει το λόγο ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω σε πόσες λεπτομέρειες πρέπει να περάσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε ότι έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη νομοθεσία όπου αναφερόμαστε στην αρχή της ε, αναλογικότητας και έχουμε και την έκθεση για την ευφύη νομοθεσία. Θα προσπαθήσω γρήγορα να καλύψω τα θέματα αυτά, με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και έχετε πάρει επίση και την έκθεση επί της οποίας εγώ γνωμοδοτώ. Όσον αφορά την αναλογικότητα και την επικουρικότητα, όσον αφορά τις δύο αυτές αρχές, θα πρέπει εδώ πέρα να υπογραμμίσουμε ότι προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ των νέων πρωτοβουλειών που προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει ότι στο μέλλον θα πρέπει σε τέσσερις κυρίως τομείς οι αρχές αυτές να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Καλύτερη νομοθεσία, μετανάστευση, καλύτερη αντιμετώπιση του καταναλωτή, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη νομοθεσία για την ενέργεια. Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα δύο θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πόσα θα πρέπει να συντονιστούν επί των τέσσερων αυτών θεμάτων, δεν πιστεύω πάντως ότι θα χρειαστεί να λώσουν πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε έπειτα και την ανακοίνωση για την ευφυή νομοθεσία που είχε ως στόχο να εξορθολογήσει την νομοθετική διαδικασία και να την κάνει πιο αποτελεσματική όσον αφορά την εσωτερική αγορά, προσβλέποντας σε μια βελτίωση τη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά προκειμένου όλο και περισσότεροι παράγοντε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν. Λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προχωρήσει σε οκτώ νέες πρωτοβουλίες και έχουμε και την πολύ σημαντική αυτή νέα πρωτοβουλία για το ότι ε, οποιαδήποτε νέα νομοθεσία θα πρέπει να υπόκειται σε μια πολύ καλύτερη αξιολόγηση από αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Πάλι η μεγαλύτερη πρόσβαση είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει πάρα πολύ σε αυτό, στην ποιοτική αξιολόγηση επίσης και θέλει να μειωθεί το 2012, και αυτό ακούγεται ιδιαίτερα φιλόδοξο, το γραφειοκρατικό άχθος. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να βελτιωθούν οι ε, ιστοσελίδες ε, που ε, προβλέπονται στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς για την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και για οποιαδήποτε πιθανότητα προσφυγής. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα ήθελα εγώ να θίξω και τα σημεία τα οποία συζητά και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων με τον εισηγητή της εκεί. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα οποία βλέπετε στην γνωμοδότηση ή μάλλον θα δείτε στην γνωμοδότηση την οποία θα διανύμω στα μέλη της Επιτροπής. Όσον αφορά την, την αξιολόγηση αντικτύπου, θεωρώ ότι ε, θα αποτελούσε βελτίωση το να έχουμε μια πιο ενισχυμένη αξιολόγηση Προτού ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία, αλλά αυτό που έχουμε δει πολλές φορές είναι ότι ε, υπάρχουν πολλέ τροποποιήσει που ε, υποβάλλονται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και που ουσιαστικά τροποποιούν σημαντικά την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία στην αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου να μπορούμε να επικαιροποιούμε, να ενημερώνουμε τι μελέτε αυτέ αντικτύπου κάθε φορά που προβλέπονται τροποποιήσει από τα θεσμικά όργανα. Δεύτερον, έγινε μία πρόταση από τα Εθνικά Κοινοβούλια να βελτιωθεί το, η ιστοσελίδα LEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUR LEX. Προβλέπεται αυτό στην έκθεση και θα συμπεριληφθεί και στη δικιά μου την γνωμοδότηση. Τρίτον, ακούστηκαν κάποια παράπονα για το ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου ουσιαστικά περιλαμβάνουν κάποια ακαθάριστα αριθμητικά, αριθμητικά στοιχεία και δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο ελήψη καθαρών αριθμητικών στοιχείων να ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος από οικονομικής πλευράς. Προβλέπω να το υποβάλουμε το ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τροποποιήσει την πολιτική που ακολουθεί στο μέλλον. Τέταρτον, στην έκθεση φαίνεται ότι το πρόγραμμα μείωσης του διοικητικού άχθους θα λειτουργήσει μέχρι το 2012. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι μέχρι τα τέλη του 2012 θα έχουμε ε, επιτύχει τους στόχους αυτούς και είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον και να μην ολοκληρωθεί το 2012. Προτείνω να έχουμε μια ρεαλιστική αξιολόγηση του αν μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέχρι το 2012 και τι θα γίνει στη συνέχεια μετά το 2012. Είναι σημαντικό να μην σταματήσει τη διαδικασία. Πέμπτον, και ολοκληρώνω, θα Ήθελα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα που έχουν εντοπίσει πολλά κράτη-μέλη αλλά και πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει με τη διαφορά εφαρμογής των κανονισμών ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης. Όχι μόνο στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, αλλά την πραγματική εφαρμογή τη στην πράξη που οδηγεί πραγματικά προβλήματα σε πάρα πολλού παράγοντε στην εσωτερική αγορά. Αναφέρθηκα στα σημαντικότερα σημεία στα οποία έχει επιμείνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, τα σημεία τα οποία θα συμπεριλάβω εγώ στη δικιά μου την γνωμοδότηση. Θα διανεμηθεί η γνωμοδότησή μου αυτή σε όλα τα μέλη τη επιτροπή μα, καθώ επίση και στην γραμματεία της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων και ελπίζω να καταφέρουμε να κινηθούμε γρήγορα έτσι ώστε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να μπορέσει να λάβει την δική μα την γνωμοδότηση και να μπορέσει να ψηφίσει την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Ιουνίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μέσσερ Σμιτ. Ο κύριος Γκερέρο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μέσσερ Σμιτ. Ο σκιώδης συζητής μας, ο κύριος Βιτάλ Μορέιρα, θα επιθυμούσε να παρευρίσκεται σήμερα εδώ και να σας εξηγήσει προσωπικά, να σας παρουσιάσει τις θέσεις τους. Αλλά επειδή τελευταία στιγμή μπήκε αυτό το θέμα στην ημερήσια διαταξή και είχε άλλη ανηλυμένη υποχρέωση προηγουμένως, ε, μου ανέθεσε να σας υποβάλω μερικές από τις δικές μας θέσεις και προτάσεις. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό. Αξίζει την προσοχή μας. Κάθε χρόνο μας απασχολεί. και μπορούμε να ε, στείλουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τη γνωμοδότησή μας. Είναι γεγονός όλο και περισσότερο αποδεκτό και παραδεκτό ότι η καλή νομοθεσία δεν είναι απλώς ένα νομικό θέμα, αλλά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που συνδέεται πάρα πολύ με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη όλο και περισσότερο το θετή είναι σημαντικό για την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας και του συστήματος γενικά. Ωραία. Τούτων λεχθέντων. Ποια είναι η αφετηρία μας. Ε, πώς θα αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση, το υπερβολικό βάρος ε, και πώς μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και τα άχρηστα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια. Όλο και περισσότερο έχουμε τέτοια προβλήματα και προσκόμματα που δεν είναι απαραίτητα για τη νομική ε, δουλειά. Λοιπόν, μείωση των διοικητικών εμποδίων, απλούστευση, χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπου ε, μπορεί να γίνει αυτό, να επεκταθεί. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Μέσερ Σμιτ, έξυπνη ευφυής ρύθμιση είναι κάτι που αφορά όλα τα πεδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οικονομικά προγράμματα. Και δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι αυτό το θέμα το οικονομικό ενδιαφέρει σήμερα όλη την Ένωση και το Κοινοβούλιο όλος ιδιαίτερος. Θα πρέπει όλο και περισσότερο να προβλέπουμε τον αντίκτυπο που θα έχει μια ρύθμιση, εξάντε δηλαδή η εκτίμηση του τι θα σημάνει αυτό και εξπόστο όμως, εκ των υστέρων να δούμε πώς λειτουργήσε, πώς μεταφράστηκε, εφαρμόστηκε στην πράξη, ε, να διορθωθούν ε, κάποιες ε, αποκλήσεις, παρεκκλήσεις και να δούμε τι λειτουργήσε καλά και να διευρύνουμε την επιτυχία. Λοιπόν, εκτίμηση εκ των πρώτων, αξιολόγηση εκ των υστέρων. Και τέλος, για να πούμε και νομοθέτες εμείς πλέον με το Συμβούλιο, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, είμαστε υποχρεωμένοι να νομοθετούμε κοντά στο πολίτη με τρόπο διαφανή και εύληπτο για το σύνολο της κοινωνίας. Και δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά λεπτομερής, σχολαστική, τεχνική η νομοθεσία, υπερβολικά... Ε, ακριβώς σχολαστική, γιατί ε, έχουμε το τελικό πολιτικό έλεγχο στις κατεξουσιοδότηση πράξης και δεν θα πρέπει να έχουμε τόση αγωνία και να ορίζουμε μέχρι και τελευταία τελεία ε, σημείο προς σημείο κάθε νομοθεσία. Να είναι πιο κοντά στον πολίτη, πιο απλή νομοθεσία και πιο διάφανη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μέσσερ Σμιτ θέλει να απαντήσει στην παρέμβαση του κύριου Γκερέρο. Δεν έχουμε κάποιον άλλον που να ζητά τον λόγο. Νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε επί του θέματος. Όλοι θέλουμε ο κανονισμός για την εσωτερική αγορά να λειτουργήσει ομαλά, και να εφαρμοστεί όσο πιο απλά για τους ενδιαφερομένους. Σημείωσα τις προτάσεις σας και τις απόψεις σας και θα τις συμπεριλάβω στο σχέδιο κειμένου που θα σας διανεμηθεί και μετά ο κύριος ε, Βιτάλ Μοραέια ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να κάνει περαιτέρω προτάσεις ε, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημείο αυτό. Ο συνάδελφος Μέσερ Σμιτ ε, σας είπε ήδη ότι θα σας διανεμηθεί η γνωμοδότησή του. Δεν θα παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση, επομένως κατάθεση τροπολογιών, αν συμφωνείτε, 20, μέχρι τις 24 Μαΐου. Πέρασε συνεδρία της Επιτροπής λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9. θα έχουμε και την κρόαση του συναδέλφου Σάγερ για το Ουγγρικό Σύνταγμα, όπως μας είπε η συνάδελφος ε, Ουργάη σήμερα. Και τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για την ε, συνεδρίαση των συντονιστών, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως και να κάνουμε το εξή αν συμφωνείτε. Να ξεκινήσουμε την εξέταση των ε, ποιον, το πιο σημαντικών θεμάτων, τα κατεπήγοντα και να κάνουμε αύριο την υπόλοιπη συνεδρία των συντονιστών διότι νομίζω ότι η αυριανή μέρα θα είναι αρκετά σύντομη και θα μας ε, δώσει κάποιο επιπλέον χρόνο για να κάνουμε την συνεδρία των συντονιστών αύριο.